Das verantwortliche Mitglied des Rechnungshofs ist ebenfalls unter uns. Herzlich willkommen. Έχουμε εκπρόσωπο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, θα τον ε, καλωσορίσουμε. Θα δώσουμε τώρα, θα δούμε ποιος θα πάρει το λόγο. Θα αρχίσει ο κύριος Πυρίνσκι με την εισαγωγή. Λοιπόν, πέρα, αρχίστε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησε αυτή η ακρόση οφείλεται ε, στα προνόμια που έχει η Επιτροπή στα πλαίσια του κανονισμού των κοινών διατάξεων, άρθρο 58, τους πόρους δηλαδή που έχει η, στη διάθεση της Επιτροπή και την ε, πρόσθετη πρωτοβουλία που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να παράσχει πρόσθετη βοήθεια στα κράτη-μέλη για να μπορέσει να ενισχυθεί η δυνατότητά τους να απορροφήσουν ε, με σωστό τρόπο τα κονδύλια και επίσης ε, τα ποσά που διατίθενται από τα προενταξιακά ταμεία στις υποψηφίες χώρες. Για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της χώρας και για την απαλλαγή από τον προπολογισμό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει από την Κομισιόν να προσφέρει περισσότερη τεχνική βοήθεια στα κράτη-μέλη και να διευκολύνει τι βέλτιστε πρακτικέ όπου υπάρχουν για την καλύτερη ε, ε, χρήση των ε, κονδυλίων. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στη ετήσια εκθεσή του και σε άλλε περιπτώσει έχει εκδώσει συστάσεις γι' αυτό το λόγο και θα πρέπει με αυτή την ευκαιρία να έχουν τη δυνατότητα οι εμπλεκόμενοι να εκφράσουν απόψεις σχετικά με την εφαρμογή της υποχρέωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βοηθήσει τα κράτη-μέλη για τη χρήση των κονδυλίων και να πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα. Η Επιτροπή και το ε, Δικαστήριο φυσικά θα, δώσουν, ε, θα εκφράσουν θέσεις ε, και απόψεις. Πιστεύω ότι ο τίτλος της ακρόασης εκφράζει τους βασικούς στόχους που πρέπει να επιδιωχθούν. Δηλαδή, καταρχήν, η προσπάθεια να εντοπιστούν τα διάφορα προβλήματα των κρατών μελών που έχουν σχέση με την ορθή απορρόφηση των κονδυλίων και δεύτερον να ε, διατυπωθούν λύσεις και την, προοπτική του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να βοηθήσει τα κονδύλια, να... τις χώρες να απορροφήσουν σωστά τα κονδύλια. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι σήμερα έχουμε κάθε λόγο να εξετάσουμε με σοβαρότητα το, τα θέματα αυτά, δεδομένου ότι η εφαρμογή της πολιτικής συνοχής στην παρούσα προγραμματική περίοδο μοιάζει να καθυστερεί και άρα δημιουργούνται ανησυχίες από τα μέσα της φετινής χρονιάς τα ποσά που έχουν δαπανηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο των διαρθρωτικών κονδυλίων είναι 27,7% και οι δαπάνες είναι σχεδόν 3,2% σε σύγκριση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο του 2009, το τρίτο χρόνο δηλαδή της περίοδου, η κατάσταση διαφέρει. Τα, ήταν 40,5% και οι δαπάνε ήταν 12,6%. Δηλαδή έχουμε διπλάσια ή τριπλάσια ποσά ε, κατά την προηγούμενη περίοδο σε σχέση με την παρούσα, πράγμα που μάλλον θα έπρεπε να σημαίνει το αντίστροφο. Φυσικά υπάρχει μεγάλη διάσταση ε, από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Κυρίως στον τομέα των δαπανών υπάρχουν οι εξαιρετικές επιδόσεις, Λιθουανία, Ελλάδα, Πορτογαλία που έχουν ε, πετύχει το 7 ή και 8% ενώ η Αυστραλία, Ορλανδία και, η Αυστρία, Ορλανδία και Ρουμανία έχουν πολύ χαμηλές επιδόσεις. Ε, ένα άλλο θέμα που είναι περίεργο το, ποσό, το, ο ρυθμός σε σχέση με τις προγνώσεις, τις αρχικές προγνώσεις για τις αιτήσει πληρωμής. Το 2016 ήταν μόνο 46% των ε, πραγματικών ε, αιτήσεων που είχαν υποβληθεί ε, σε σχέση με τα προβλεπόμενα ποσά της χρονιάς. Το χαμηλότερο είναι, προέρχονται από χώρες Ολλανδία, Ρουμανία και Κροανία και τα υψηλότερα από τη Σουηδία 194%, Φιλανδία και Πολωνία. Οπότε δεν θέλω να επισέλθω στα αίτια τη στιγμή αυτή. Ενδεχομένως ο καθένας μας να έχει ε, δικές του ε, ιδέες για τα αίτια. Έχουν συνταχθεί και ειδικέ εκθέσεις, έχει συζητηθεί και στο ελεγκτικό συνέδριο το θέμα αυτό επανειλημμένος, με διάφορες, σε διάφορες συνθέσεις. Δεν θέλω να τα ε, ανακεφαλαιώσω όλα αυτά, ούτε... Ε, εξάλλου πρέπει να περιμένουμε τους ε, μιλητές που θα ακολουθήσουν. Θα ήθελα όμως τη στιγμή αυτή να επισύρω την προσοχή σας σε ένα κεντρικό έβριμα. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να το προσέξουμε. Έγινε το Μάρτιο του 2014 μια ανακοίνωση κομισιών από την προηγούμενη Επιτροπή που κατέληγε στο ανησυχητικό συμπέρασμα ότι η λεγόμενη ε, ε, ο λεγόμενος μηχανισμός σύγκλησης που είχε ε, ε, υλοποιηθεί με επιτυχία μέχρι το 2008, μέχρι την κρίση από την Κομισιόν, είχε καθυστερήσει και ενδεχομένως οπισθοδρομούσε. Αυτό το έβριμα περιλαμβάνεται και στο έγγραφο περισυλλογής για την κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο υπέβαλε η Κομισιόν πριν από δύο μήνες. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, εν μέσω της τρίτης χρονιάς της τρέχουσας περίοδου συνοχής βρισκόμαστε στην ίδια εξαιρετικά ανησυχητική κατάσταση. Δηλαδή η πολιτική συνοχής όχι μόνο δεν ε, αυξάνει την, ε, το ρυθμό της, αλλά βρίσκεται σε μια καθόλου ικανοποιητική κατάσταση και σε μερικές περιπτώσεις υπάρχουν σημαντικοί δείκτες που δείχνουν ότι η συνοχή προχωρεί αρνητικά. Μιλάμε για αποσυνοχή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και προσβλέπω στην πολύ σημαντική αυτή συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σωστά ε, ε, ε, καλούμαστε να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ για τις μεγάλες προσπάθειές σα. Το λόγο θα δώσω στον κύριο Ντορέιτ από το ελεγκτικό συνέδριο. Χαίρομαι που είστε μαζί μας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πρέπει να ομολογήσω ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εργάζεται επί μια ειδική έκθεσης για την απορρόφηση των κονδυλίων και θα εκδώσουμε την έκθεσή μας ε, στα τέλη του Φεβρουαρίου του χρόνου. Δεν μπορώ λοιπόν να σας δώσω τώρα κάποια ενημέρωση για τις συστάσεις ή για τα συμπεράσματά μας. Απλώς θα σας πω κάποιες ιδέες. Το κύριο, το κύριο πόρισμα της εκθεσής μας θα είναι ότι συστημικά προβλήματα πρόφησης έχουν παρατηρηθεί από το 2000 η απορρόφηση των κονδυλίων ξεκινάει αργά στην αρχή της προγραμματικής ε, περίοδου και στο έγγραφο που εκδόθηκε από την πλευρά σας για τα διδάγματα από το κλείσιμο του προγράμματος θα δείτε που είναι τα προβλήματα. Το μοντέλο το δεν ε, έχει αλλάξει μετά την ε, διεύρυνση. Περίπου το 30% των ε, κονδυλίων πληρώνονται μετά το τέλος της προγραμματικής περίοδου και για την ε, περίοδο 2007-2013 οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων έπρεπε να δαπανηθούν ε, μετά από 2-3 χρόνια. Ο κανόνας νη συν 2. Ο κανόνας αυτός δεν έχει ε, κάποια επιρροή ε, κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περίοδου, όμως αυτά τα μέτρα έχουν περιορίσει τις ε, πληρωμές ε, για ένα χρονικό διάστημα μετά το τέλος της περίοδου εδώ βλέπετε πως, ότι δεν αλλάζει το μοντέλο απορρόφησης για το ΕΤΠΑ. Υπάρχει μία απόκληση για τα ποσά που έχουν δεσμευτεί και αυτά που πληρώθηκαν. Βλέπετε ότι παρά τις αλλαγές στους νομικούς κανονισμούς, το μοντέλο της δαπάνης ε, παραμένει παρόμοιο. Τα μοντέλα διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών. Και αυτό ισχύει για το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ισχύει και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όπως είδατε στην προηγούμενη διαφάνεια. Η απορρόφηση του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την περίοδο 2000-2006 είναι της περίοδου 2007-2013 γίνονται δέσμευση των πιστώσεων για 7 χρόνια και μετά από 7 χρόνια μόνο το 70% των δεσμευμένων πιστώσεων ε, έχουν δαπανηθεί. Χρειάζονται περίπου 10 χρόνια για να δαπανηθούν τα κατανοημένα χρήματα. Το ίδιο ισχύει για το κοινωνικό ταμείο βλέπετε εδώ παρόμοια καμπύλη μεταξύ διάφορων κονδυλίων και περιόδους και τα ίδια σχόλια ισχύουν και για το γράφημα αυτό όπως και για το προηγούμενο. Πριν τον κανόνα 2, δηλαδή μεταξύ 2000 και 2006, οι πληρωμές συνέχισαν για πολλά χρόνια μετά την προγραμματική περίοδο. Ο κανόνας νησιν 2 εισήγαγε το ε, περίοδο 2007-2013 ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα όπου τα δεσμευμένα ποσά μπορούν να δαπανηθούν. Πριν την εισαγωγή αυτού του κανόνα για την προγραμματική περίοδο 2000-2006 συνεχίστηκε μέχρι το 2013 συνεχίστηκαν οι πληρωμές. Πιθανά συμπεράσματα. Καταρχήν, η Κομισιόν ενέκρινε το κανονιστικό πλαίσιο και τα επιχειρησιακά προγράμματα πολύ αργά. Η επικάλυψη του πολιτού στο μεσονομικού πλασίου είναι ε, ουσιαστικά πηγή προβλημάτων. Παρακαλώ να δείτε την ε, έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου για το κλείσιμο των προγραμμάτων. Πολύ συχνά τα κράτη-μέλη κάνουν ταυτόχρονα προσπάθειες να κλείσουν το παλιό πρόγραμμα και να ξανανοίξουν να ανοίξουν το καινούριο. Τα Κομισιόν και τα κράτη-μέλη ανείχνευσαν πολύ αργά την εργή απορρόφηση. Τα προβλήματα με την απορρόφηση εντοπίστηκαν καταρχήν σε επίπεδο κρατών μελών, αλλά θα μπορούσαν να έχουν εντοπιστεί και νωρίτερα. Παρά την ύπαρξη πολλών εργαλείων υποβολής εκθέσεων για την ε, ετήσια εφαρμογή, δεν χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα εργαλεία για την αποτροπή των προβλημάτων. Πολλά μέτρα που προτίθηκαν από την Κομισιόν εφαρμόστηκαν από τα κράτη-μέλη για τη βελτίωση της ε, απορρόφησης επικεντρώθηκαν λιγότερο στις επιδόσεις. Τα κράτη-μέλη και κομισιόν ανέλαβαν συγκεκριμένες ε, πρωτοβουλίες δημιουργήσαν μία task force για την ε, βελτίωση του ποσοστού απορρόφησης. Τα περισσότερα μέτρα ε, που βουλεύτησαν από τα κράτη-μέλη προβλέπονται στην ομοθεσία. Η χρηματοοικονομική μηχανική μπορεί να οδηγήσει ώστε να επιληθούν ε, κάποια προβλήματα για την περίοδο 2014-2020. Ο παραπρογραμματισμός είναι το πιο σημαντικό μέτρο, όμως πρέπει να αναθεωρηθεί και η λογική της ε, παρέμβασης. Μερικές φορές ε, χρειάζεται να γίνει νέα ανακατανομή των κονδυλίων, όμως αυτό πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους ε, του επιχειρηματικού προγράμματος ή του κράτους μέλους. Δεν θα πρέπει η έμφαση στην απορρόφηση να αντικαταστήσει την προσπάθεια να έχουμε υγιή οικονομική διαχείριση και συμμόρφωση και να πάμε στις πιθανές συστάσεις η Κομισιόν ε, πρέπει να προσαρμόσει το πλαίσιο της νομοθεσίας της για να εξαλείψει τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την επικάλυψη της προγραμματικής περίοδου. Η Κομισιόν θα πρέπει να εγκρίνει τα προγράμματα και τους κανονισμούς εγκαίρους. Το πρόβλημα των περιόδων επικάλυψης θα χρειαστεί να γίνει προσαρμογή μακροπρόθεσμου οικονομικού σχεδιασμού. Μία λύση θα ήταν να ξεκινήσει με ένα προγραμματική περίοδο το 2022 και περίοδος 2020-2022 να φεθεί για το κλείσιμο του προγράμματος και να είναι προπροσκευαστική για το επόμενο. Επίσης, η Κομισιόν θα πρέπει να περιορίσει ε, την χρήση των καταναμημένων πόρων μετά το τέλος ε, της ε, προγραμματικής περίοδου μέχρι δύο χρόνια μετά το τέλος της περίοδου και τρία χρόνια σε ειδική περίπτωση. Η Κομισιόν θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει ε, τακτική υποβολή εκθέσεων και παρακολούθηση για διορθωτικές δράσεις εγκαίρως. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν καλύτερες εκθέσεις και να προβλέπουν τα προβλήματα. Θα πρέπει να εισαχθεί υποβολή εκθέσεων ε, και να συνοδεύει τις αιτήσιες ε, υποβολές εκθέσεων πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα καθήκοντα ω μέρο ευρύτερη στρατηγική. Πολλά θέματα σχετίζονται με την δικατική ικανότητα του κρατου μέλους. Η Κομισιόν θα πρέπει να, να υιοθετήσει πράξεις για να ενισχύσει την ικανότητα των, κρατών, των κρατών μελών να διαχειρίζονται και να εφαρμόζουν τα διευθυντικά ταμεία. Επίση, η Κομισιόν θα πρέπει να προσαρμόσει του στόχου και του δείκτε σύμφωνα με την λογική παρέμβαση να αλλάξουν τα προγράμματα τα επιχειρησιακά. Θα... Η εστίαση στις επιδόσεις θα πρέπει να είναι η κυρία προτεραιότητα. οποιοδήποτε επαναπρογραμματισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει αναθεώρηση της λογικής παρέμβασης. Η Κομισιόν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει στα δεδομένα απορρόφησης μόνο τα ποσά που έχουν ε, αποδεσμευτεί και όχι ε, ποσά που δεν έχουν δαπανηθεί έτσι λοιπόν δεν, ε, αυτό το αυτό το θέμα έχει επιληθεί στη νέα προγραμματική περίοδο. Αυτά, Πρόεδρε, είναι τα δικά μας σχόλια για την έκθεση που θα εκδώσουμε του χρόνου του Φεβρουάριου. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε την έκθεση σίγουρα. Αλλά τι περιέχει τέλος πάντων. Ε, υπάρχει κάποιος ε, που είναι από την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ για τα περιφερειακά ζητήματα για να μας ε, μιλήσει, ναι ή όχι. Είστε εδώ κάποιος. Also, ja. Naja, ich war να ανησυχώ λίγο. Ναι. Εντάξει, θα τα καταφέρουμε. Με ακούτε? Όταν μπορείτε, παρακαλώ, να πάρετε το λόγο. Καλώς ήρθατε. Ωραία. Μπορείτε τώρα να είστε, ναι. Ε, ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, ε, άργησα, αλλά οι Βρυξέλλες πρέπει να μπουν στις καινοτόμε δράσεις για τις μεταφορές. Δεν υπάρχει ούτε καινοτομία, ούτε ασφάλεια. Ε, δέκα λεπτά χρειάστηκε για να μπω, συγγνώμη που το λέω, αλλά τέλος πάντων. Στην περίοδο 2017-2013 Υπάρχει ε, ο σχετικός έλεγχος ε, από την αρμόδια γενική διεύθυνση. Έχουμε λάβει τις εκθέσεις κληθήματος ε, από τα κράτη-μέλη τέλη Μαρτίου ήταν η προθεσμία και είχαμε πέντε μήνες στην Κομισιόν να τα εξετάσουμε γιατί υπήρχαν πολλά πράγματα που πρέπει να τα μελετήσουμε. Μπορώ πάντως να σας πω ότι σε ό,τι αφορά ε, το πρόγραμμα αυτό για το Γιβραλτάρ καταρχάς. Ε, πάνω από 20 παρατηρήσεις έχουμε για το κλείσουμε αυτό. Άρα έχουμε τα πρώτα στοιχεία που λένε ότι κλείνουν ε, τα προγράμματα, αλλά θα χρειαστεί λίγο παραπάνω χρόνος για να γίνει σωστά και οριστικά το κλείσιμο. Επίσης, ταυτόχρονα, Κάνουμε και την ε, των αξιολόγηση για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής και με τα χαράς μπορούμε να σας πούμε ότι είχαμε επιστροφή επενδύσεων πολύ θετική για κάθε ευρώ σχεδόν 3 ευρώ. Δεν είναι ένα χρηματοπιστωτικό μέσο, βέβαια. Στην περίοδο 7-13 κάθε περιφέρεια στην Ευρώπη υποφελήθηκε από αυτά τα κονδύλια. 4,2% το ΑΕΠ είναι για τις χώρες συνοχής και ακόμη και σε άλλες χώρες, ε, όχι συνοχής, ε, κάτω είναι 0,4 και πάλι είναι σημαντικός ο αντίκτυπος για την οικονομική ανάπτυξη, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά σε αυτή την περίοδο ε, δήλθαν μεγάλη κρίση περιφέρειας και χωρίς ε, την υποστήριξη από τα κονδύλια αυτά θα είχαν υποφέρει πολύ περισσότερο. Η καταρακτική ανάλυση αυτών των ε, πέσεων κλεισίματο προσπαθούνται να βρούμε ακόμα <clears throat> τις σωστές τιμέ και αξίε, αλλά τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι σε 400.000 μικρομεσαίε επιχειρήσεις έχουν λάβει υποστήριξη και εξ αυτών 120.000 ήταν νεοφύς επιχειρήσεις, άρα δημιουργήθηκαν νέε θέσει εργασία παρά την κρίση και το πώς επηρέασε πολλές από αυτές τις περιφέρειες. Επίσης υποστηρίξαμε την έρευνα και την καινοτομία για τις νέες τεχνολογίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Ένα ακόμα δύο εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν 3 εκατομμύρια όμως είναι καθαρά συνολικά αυτές οι θέσεις. Υπάρχουν σημαντικές συμφορήσεις βέβαια όπως καταλαβαίνετε σε δίκτυα για τα, διευρωπαϊκά, τα δίκτυα μεταφορών δίνεται πολύ υποστήριξη. 6.000 ε, χιλιόμετρα οδικού δικτύου και η κινητικότητα υποστηρίζεται. τα μέτρο, το πραστιακό, τη διασύνδεση των αστικών περιοχών με τα περίχωρα κτλ. Και με το Ταμείο Συνεχίσης συνεχίζουμε να επενδύουμε σε σημαντικά για τους πολίτες ζητήματα, καθαρό πόσιμο νερό και επεξεργασία λιμάτων. Συνεχίζουμε και σε αυτήν την περίοδο. Επίσης, ξεκινήσαμε ήδη ε, να εργαζόμαστε για την ψηφιακή Ευρώπη. 15 εκατομμύρια πολίτες έχουν πλέον πρόσβαση σε νέα ή βελτιωμένα ευρυζωνικά δίκτυα. Όπως είπα, την τελική εικόνα θα την έχουμε όταν ολοκληρωθεί η εικόνα αυτή, ε, ή μάλλον συγγνώμη για διαδικασια των κλεισιμάτων. Μάλλον τον Οκτώβριο δηλαδή θα έχουμε πιο ακριβή στοιχεία. Αυτό που θέλω να πω βέβαια, διότι αυτό το θέμα είναι lessons learned, δηλαδή τι δάγματα αντλήσαμε για την περίοδο, για να τα εκμεταλλευτούμε για την περίοδο την επόμενη. Για την επόμενη περίοδο έχουμε ενσωματώσει πολλά από αυτά που ήταν στην περίοδο 7-13. Είχαμε ελέγχου επιδόσεων από το Ελληνικό Συνέδριο, συζητάτε εδώ στο Κοινοβούλιο, συζητάτε και το θέμα συζητείται και στα κρατημέλη. Εμείς Εμεί εστιάζουμε στην καλύτερη ε, των πόρων, στι καλύτερε δαπάνε. Εδώ για, για τη νέα περίοδο 14-20. Τα νέα στοιχεία που θα συνεισφέρουν και ήδη συνεισφέρουν στην πιο αποτελεσματική των κονδυλίων είναι φυσικά οι αιρεσιμότητε οι εξάντερες ημότητες. Φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν στρατηγικοί στόχοι για τι επενδύσεις, ώστε να φαίνεται ότι εντάσσονται οι ε, στις, ε, στους αναπτυξιακού στόχους. Υπάρχουν και κάποια άλλα, υπάρχουν οριζόντια στοιχεία όπως είναι διαγωνισμοί και υπάρχουν και κάποια τομεακά. Στις μεταφορές κατά χάρη είδαμε ότι πολλέ περιφέρειες και πολλά κρατημέλη δεν είχαν γενικά σχέδια Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι η στρατηγική για την ευφύ εξειδίκευση ως εξαντέρεσιμότητα. Για την και την καινοτομία. Στο Ελσίνκι ήμασταν πριν και προσπαθήσαμε να μελετήσουμε εκεί τα στοιχεία. Και είναι προφανές ότι οι χώρες που μένουν πίσω, μου ε, ενεκτούν, με την ευφύ εξειδίκευση μπορούν να, να στοχεύσουν καλύτερα στις επενδύσεις, ξέρουν καλύτερα τι να κάνουν και υπάρχει και διάλογο μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων φόρων που βελτιώνεται και αυτό είναι πολύ καλό. Αυτή η προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Η ευφύ εξειδικευσή. Κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον είναι ότι οι πιο ανεπτυγμένε περιφέρειε, ε, είχαμε μια παρουσία από την Αυστρία ε, γύρω στη Βιέννη, που έλεγαν ότι πλέον υπάρχει μια ενιαία διαδικασία και στρατηγική για την ευφύ εξειδίκευση. Σε ό,τι διαφορά το πλαίσιο επιπτώσεων, πλέον είναι σαφές και περιλαμβάνονται πλέον σαφείς δείκτες για να βελτιώσουν τους αντικτύπους. Και είχαμε εδώ νομίζω τη συζήτηση ήδη στο παρελθόν τα πράγματα δεν είναι τέλεια, θα πρέπει να εξορθολογήσουμε τους δείκτες μεταξύ των ταμείων, θα πρέπει να φροντίσουμε ότι περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα να μην αλλάξει τη μέση, αλλά να αποδώσει. Και γι' αυτό συνεχίζουμε το έργο μας και παρακολουθούμε εκ του και στην κατάσταση, για να δούμε πώς αυτό το, αυτό το πλαίσιο επιδόσεων προχωρά και βέβαια και το 6% του αποθεματικού που θα διανεμηθεί αργότερα. Επίσης έχουμε και άμεση ενδιαφέρον από τις πόλεις που ήταν και το ζητούμενο. Υπάρχουν πόλεις που έχουν σωματωμένες στρατηγικές. Θέλαμε να δημιουργήσουμε λειτουργικές περιοχές και τον ε, Σεπτέμβριο θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ε, μελέτη για το πώς ε, πόσο ενδιαφέρον υπάρχει. Μπορεί να καθυστέρησε η αρχή αυτή γιατί ήταν κάτι καινούργιο, αλλά βλέπουμε ότι παρόλα αυτά υπάρχει ενδιαφέρον από όλη την Ευρώπη. Άρα θα προωθηθεί η συνεργασία, η ολοκλήρωση και μια ολιστική προσέγγιση. Και το ενσύκι μας ευχαρίστησε. Γιατί λέω ότι πριν κάπως ήταν κατακαιρματισμένοι διάσπαρτοι και τώρα ε, κοιτάνε όλη ε, την ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση. Για αυτή την περίοδο 14-20 πράγματα, ποσοστά απορρόφησης, εκτιμήσεις δεν και τόσο. Ε, θετικές όσο θα περιμέναμε και για φέτος όμως η επιλογή των διαφόρων ε, ενεργειών ε, αυξάνεται. 180 δις ήδη επενδύονται επί τόπου με όλες αυτές τις νέες, με τους νέους όρους και προϋποθέσεις για να είναι πιο στοχευμένες οι επενδύσεις. Αυτό που μάθαμε από την περίοδο 7-13 είναι ότι θα πρέπει να εργάζεται προορατικά η Κομισιόν μαζί με πολλά κράτη και πολλές περιφέρειες. Κάναμε ό,τι μπορούμε για να δούμε τι προβλήματα ε, δημιουργούν οι περίεργες κατευθυντήριες γραμμές και να υπάρξει ε, βελτίωση ήδη από τα τέλη αυτής της περίοδου, αλλά για την επόμενη τα αιτία θα συνεχίσουμε έτσι να δουλεύουμε. Έχουμε το Unit Better Implementation και συνεργαζόμαστε και με τα κράτη-μέλη. Μόλις ε, επέστρεψα από το Quest και χαίρομαι που βλέπω εδώ τη Μικαέλα, γιατί από κοινού σχεδιάσαμε το σχέδιο δράσης το οποίο εφαρμοστεί για να αποφύγουμε συμφορήσεις ε, στην απορρόφηση και ε, decommitments, αποδεσμεύσεις. Η χώρα αυτή έχει πολλά ποσά που παίρνει. Με τις υπολοιπόμες περιοχές έχουμε πιλωτικά στην Πολωνία για παράδειγμα για να υπάρξει σχέτιση με την επιλογή προγραμμάτων στο πλαίσιο της εφίους Εξειδίκευση Στη Ρουμανία κάνουν το ίδιο. Επίση έχουμε πλέον ένα ειδικό σύστημα παρακολούθησης που βλέπουμε τις αιτήσεις εκθέσεις υλοποίησης, τις αναλύουμε και εντοπίζουμε τα προγράμματα που είναι στη χειρότερη κατάσταση. Τα έχουμε εντοπίσει, πρέπει να σας πω, και μαζί με τις διαχειριστικές αρχές φτιάχνουμε μικρά σχέδια δράσης για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να σημειώσουμε πρόοδο με την υλοποίηση, που θέλουμε βέβαια να είναι και ποιοτική. Βασική αρχή μας είναι η διαφάνεια. Υπάρχει μια πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων που επικαιροποιούμε, χωρίς να θέλουμε να κατονομάσουμε και να εκθέσουμε κανέναν. Απλά προσπαθούμε να δείξουν ότι υπάρχουν κάποιοι που τα καταφέρουν καλύτερα τα λοιπά. Τέλος, ο ορισμός, το designation, μάλλον θα ξεκινήσει σύντομα και θα περάσει και στον επόμενο, στον επόμενο γύρο, στην επόμενη πταετία. Επίσης προσπαθήσαμε την τεχνική βοηθή να τη σχεδιάσουμε με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Έχουμε το peer-to-peer, -peer, για να δούμε ποιε είναι οι πραγματικέ ανάγκε και να τι με πραγματικού εμπειρογνώμου που ξέρουν γιατί μιλάνε. Χρησιμοποιούμε και το Jaspers και το Compass, άρα την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και κάποια στιγμή ελπίζω να επανέλθουμε σε αυτό, αλλά τέλο πάντων. Αυτή τη στιγμή το Jaspers, για να σα δώσω ένα παράδειγμα, που βοηθά τα κράτη-μέλη, όχι μόνο σε μεγάλα project, αλλά και σε άλλα project. Έχουμε τριμερεί συναντήσει με Jaspers, Κομισιόν και κράτη-μέλη για να συνεργαστούμε καλύτερα, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αποδείχνουμε αποτελέσματα. Σταματάω εδώ γιατί θα μου το κόψετε το μικρόφωνο σε λίγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πραγματικά μπήκα στον πειρασμό να σας κόψω το μικρόφωνο, αλλά Δεν νομίζω ότι μιλήσατε για το θέμα για απορρόφησης. Ε μιλήσατε για, τη, για τα ταμεία συνοχής, αλλά εμείς περιμέναμε να μας μιλήσετε συγκεκριμένα για τα προβλήματα απορρόφησης ε, και για τη Ρουμανία και για άλλες χώρες. Η Ρουμανία νομίζω είναι από τις πιο προβληματικές ε, υποψήφιες. Ο κύριος ε, από το Ελληνικό Συνέδριο είπε ότι έχουμε ένα πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε από το 2000 συγκεκριμένα ότι έχουμε τα ίδια μεγέθη κάθε φορά και πάντα το ελληνικό συνέδριο κάνει τις αναφορές του και τα ίδια προβλήματα ε, βλέπουμε να ανακύπτουν και από ό,τι φαίνεται δεν έχει λυθεί το ζήτημα με διοικητικά μέτρα. Έχουμε και μια δική ελληνικού συνεδρίου που μιλάει για το κατά πόσο να ε, ε, εφαρμόζονται σωστά οι στόχοι, τη σκοπιμότητα και τα λιμάνια, θυμάμαι, ήταν ένα θέμα. Αλλά νομίζω ότι πρέπει σοβαρά πλέον να ασχοληθούμε με το θέμα. Ποια είναι η ανάλυση της ΓΑΜΑ Regionalis σε ό,τι αφορά τα προβλήματα απορρόφησης και τι κάνετε για να τα αντιμετωπίσετε αυτά τα προβλήματα απορρόφησης. Σίγουρα αναχώρα είναι διαφορετικά τα προβλήματα. Αλλά υπάρχει και στο συστημικό πρόβλημα θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε ε, όταν στη περίπτωση κάθε χώρας βλέπουμε τα project και βλέπουμε ότι σε κάποιες περιφέρειες υπάρχουν πάρα πολλοί ε, πόροι από τα διευθυντικά ταμεία για παράδειγμα. Κάποιες φορές όμως τα κονδύλια αυτά ή ε, χρησιμοποιούνται για κάτι άλλο ή απλά κάθονται εκεί. Δεν χρησιμοποιούνται. Να δώσω τώρα το λόγο όμως στον εισηγητή τον κύριο Πυρίνσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σωστό να πάρω το λόγο εγώ ή μήπως να περιμένω προς το τέλος του προγράμματος. Ε, υπάρχουν ερωτήσεις. Ερωτήσεις. Κι εγώ ένιωσα ότι ο κύριος Πόπενς δεν ήταν απόλυτα σαφής επί του αντικειμένου αυτής της ακρόασης. Σε κανένα σημείο δε, της περιγραφής δεν αναφέρεται ότι ε, μας απασχολεί μόνο η περίοδος 2007-2013. Αναφέρθηκε και εκείνος σωστά ανοιχτά στοιχεία που μας δίνουν τα στοιχεία για την τρέχουσα προγραμματική περίοδος. Και κρίμα που δεν μπόρεσε να έρθει νωρίτερα, γιατί ένα από τα θέματα που προσπάθησα εγώ να επισημάνω είναι ότι κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο είναι το, ότι το ποσοστό των πραγματοποιηθησών δαπανών είναι από ό,τι μοιάζει τρεις φορές χαμηλότερο από ό,τι κατά την προηγούμενη αντίστοιχη προγραμματική περίοδο. Ο, ίδιος, ο ίδιος την ταχύτητα εισαγωγή του ανέφερε, αν δεν κάνω λάθος, ότι η Επιτροπή, η ίδια Επιτροπή έχει, νομίζω είπε, απογοητευτεί σχετικά για την κατάσταση αυτή, αλλά από τα υπόλοιπα που μας είπε, ε, έμοιαζε πολύ ικανοποιημένη η Επιτροπή με αυτά που κάνει κάτι και ότι όλα πάνε όπως πρέπει. Οπότε ρωτάω, μήπως όπως είπατε και εσείς ε, κάνει δημόσιες σχέσεις αυτή τη στιγμή στην ακρόαση η Κομισιόν ή πραγματικά δεν έχουν ε, συνέστηση του βάθους του προβλήματος, του συστημικού προβλήματος. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες, είναι μια γενική ερώτηση που κάνω. Προτείνω επίσης ο κύριος Γκέρντενς από, το ελεγκτικό συνέδριο να στείλει στον κύριο Πόπενς τις διαφάνειές του. Γιατί ενδεχομένως θα ήθελε ο κύριος Πόπενς να ακούσει τα πολλά σοβαρά και ξεκάθαρα ε, που ανέφερε το ελεγκτικό συνέδριο. Φυσικά, κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι η απορρόφηση είναι μια προσπάθεια που πραγματοποιείται και από πλευράς Επιτροπής και από πλευράς ε, κρατών μελών και ότι πρέπει να γίνει μια πολύ ε, μεγάλη προσπάθεια και τις δύο πλευρές. Όπως είπε η Επιτροπή, ε, δεν είναι μόνο το θέμα της γνώσης, είναι θέμα και των βέλτιστων πρακτικών. Πιστεύω όμως ότι είναι υποχρέωση της Επιτροπής, σύμφωνα με την ε, CPR και το άρθρο 58 του κανονισμού αυτού, ε, ότι πρέπει να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να εμπλακούν σε ευρύτερες δραστηριότητες έτσι ώστε η απορρόφηση να μην μείνει στα τωρινά επίπεδα. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον άλλο να θέλει το λόγο. Να δώσω το λόγο στους δύο μιλητές μας, ε, Πόπινς. Α, ήθελε η κυρία Αγιάλα το λόγο, φυσικά και θα προηγηθείτε εσείς, ναι, παρακαλώ. Μια ερώτηση μόνο. Θα μιλήσω ισπανικά. Ήθελα να προσθέσω σε αυτό που είπε η εισηγητής το εξή. Αυτή τη στιγμή που έχουμε τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και παράλληλα τρέχει και το Brexit, Υπάρχει ένα θέμα που ιστορικά υπήρξε με το προβλήματος της απορρόφησης ε, των πόρων, ε, και των πρόσθετων πόρων, αλλά αυτό έχει να κάνει με την απόφαση των κρατών μελών να μην συγχρηματοδοτούν για διάφορους λόγους και να διατηρούν τα ευρωπαϊκά ταμεία, τα ευρωπαϊκά κονδύλια ως ε, ουσιαστικά μια χρηματοδότηση ασφαλείας που διαπραγματεύονται με την Κομισιόν. Εγώ θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Γκρέτεν, αλλά και τον κύριο Πόπενς κυρίω, ε, και έρχεται από την ΓΑΜΑΔΕΛΤΑ Ρίτζιο, ως ποιο σημείο τώρα, το 2017, κάποια κράτη-μέλη ακόμα προσπαθούν να απορροφήσουν, να απορροφήσουν κονδύλια με ένα κυκλικό τρόπο για να διατηρήσουν ε, πολλές φορές αυτά τα χρήματα τα οποία δεν τα επενδύουν ε, και να τα έχουν ε, ουσιαστικά ως ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Ευχαριστώ κύριος Γκρέτεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τα είπατε πολύ σωστά τα πράγματα. βάλτε το δάκτυλο από τον τύπο τον και συμφωνώ. Πρέπει κάποιες φορές να κάνουμε ανάλυση των αναγκών. Ε, και επίσης πολλές φορές υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα και κάποιες περιφέρειες δεν γνωρίζουν τι να κάνουν με τα χρήματα που έχουν στη διάθεσή τους, τι λογικό να κάνουν με αυτά τα χρήματα και νομίζω ότι για την επόμενη περίοδο θα πρέπει να το σκεφτούμε πώς μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα σχόλια μου αναφέρατε τα, τα αποτελέσματα των διμερών διαπραγματεύσεων και μπορώ να σας πω ότι πραγματικά η Κομισιόν έλαβε εγκόμπια για όλο όσα κάνουμε πριν, ε, πριν υιοθετηθεί το νομοθετικό πλαίσιο από τους συνομοθέτες. Εγώ δεν διαπραγματεύομαι τους κανονισμούς, απλώς τους εφαρμόζω και γι' αυτό ήμασταν με πρακτικό πνεύμα από την αρχή και ευχαριστώ και το ελεκτικό συνέδριο που το αναγνώρισε αυτό. Επίσης αναγνώρισε ότι η νέα προγραμματική περίοδο έχει νέα στοιχεία. Δεν είναι τέλεια, αλλά υπάρχουν νέα στοιχεία που στοχεύουν στις επενδύσεις. Και αν είναι πιο αργή από την προηγούμενη, δεν είναι επειδή δεν διαπραγματευτήκαμε. Διαπραγματευτήκαμε πολύ καλά και υιοθετήσαμε κάθε λεπτομέρεια του κανονιστικού πλαισίου. Και το ίδιο έκαναν και τα κράτη-μέλη. Γιατί έπρεπε να θέσουν την ερεσιμότητα τεξάντε, το νέο πλαίσιο και όλα τα άλλα πράγματα, όπως είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση τα οποία τελικά κάνουν πιο παιδικές τις επενδύσεις μας. Και έχει και καλύτερο αντίκτυπο. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν, ήταν συμβιβασμό και είπαμε από την αρχή. Είναι ποιότητα των επενδύσεων που μετράει. Και νομίζω ότι η Επιτροπή σας είναι σε θέση να το καταλάβει. Η απορρόφηση, ναι, βέβαια, αναλύουμε τα χρηματοοικονομικά δεδομένα και μπορώ να σας ε, διαβεβαιώσω ότι κάθε μέρα θα συζητούμε αυτά και αύριο θα αναφέρω για την εφαρμογή, για την αργή απορρόφηση, θα ζητήσουμε και από τους εμπειρογνώμονες να δώσουν το δικό τους feedback. Γιατί τώρα βλέπουμε ότι ξεκινά αργά η περίοδος, αλλά η ποιότητα θα είναι καλύτερα και ακριβώς αυτό θέλουμε. Και ακόμη και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε κάποια κράτη-μέλη, εξακολουθούμε να σημειώνουμε πρόοδο και ήδη το 10% έχει αρχίσει να επενδύεται. Υπάρχουν στοιχεία λοιπόν που δεν υποστηρίζει η ιδιαίτερη Κομισιόν όπως ο κανόνας νήσιν 3, οι πολύ υψηλέ προκαταβολές, όμως σε αυτό το κανονιστικό πλαίσιο δουλεύουμε. Υπάρχουν πράγματα που είναι πέρα από τον ε, εφαρμοστικό έλεγχο. Μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο εντό του κανονιστικού πλαισίου. Τώρα αυτό αφορά τα κράτη-μέλη που καθυστερούν, κυρίως στη Ρουμανία, την Κροατία. Έχουμε δεδομένα γιατί έφτασαν οι πληρωμές ε, τελικά το 95% για την περίοδο 2007-2013 εκτός από την Ελλάδα. Και υπάρχει μια χώρα, η Κροατία, η οποία ολοκληρώνει τώρα αυτή την περίοδο γιατί μπήκε αργότερα. Και υπάρχουν και επικαλύψεις. Κλείνει το, από τη μια η περίοδος αυτή και ε, έχουμε την έναρξη της νέας περίοδου για τις μικρές ε, κυβερνήσεις. Ξέρω ότι οι μικρές ε, χώρες δεν μπορούν στη δίκησή τους να πάρουν πολύ περισσότερους ανθρώπους. Και γι' αυτό ακριβώς το πρώτο που προτείναμε στην Επίτροπο Κρέτσου και το υιοθέτησε ήταν αυτό. χτε κλείσαμε την ομάδα απλούστευσης, γιατί ξέρουμε ότι εντό του σημερινού κανονιστικού πλαισίου υπάρχουν δυνατότητες να υπάρχει μεγαλύτερη απλούστευση των ταμείων. Υπάρχει κάποιο ιστορικό, αλλά σας διαβεβαιώ, τον Οκτώβριο θα έχουμε ένα εργαστήρι και ουσιαστικά θα δούμε ε, ποιες είναι οι απλοποιημένες επιλογές του κόστους, όμως πρέπει να δείξουμε ποια είναι τα καλά παραδείγματα, όπως μας τις πρότεινε η ομάδα πλούστευσης. Υπάρχει και ένα όμνιμπους, συγκεκριμένα πράγματα θα βελτιώσουμε για τα οικονομικά μέσα, τα πλουστευμένα κόστη. Έτσι λοιπόν, συνεχώς σκεφτόμαστε τι να βελτιώσουμε. Και αν εγκρίθηκε το omnibus, διότι δεν είναι ακόμη στο Κοινοβούλιο, νομίζω ότι θα συνεισφέρει πάρα πολύ στην εφαρμογή αυτής της περίοδου. Γιατί κάποια από τα θέματα που εντοπίσαμε και μέσω της εφαρμογή και πρέπει να διορθωθούν, αυτό μπορεί να γίνει. Επίσης, είμαστε πολύ ενεργοί, συνεργαζόμαστε και με γάμα δέλτα, κάθε εβδομάδα έχουμε συναντήσεις συντονιστών, ε, μόνο από κοινού ερμηνεύουμε το κανονιστικό πλαίσιο ε, μία φορά το μήνα συναντώ του συναδέλφου από τι άλλε γενικέ διευθύνσει και συζητάμε πολλά προβλήματα. Γιατί και άλλα πρέπει να γίνουν. Συζητάμε και τι θα γίνει μετά το 2020. Όμω δεν ισχύει ότι δεν είναι προδραστική η Κομισιόν. Είμαστε ιδιαίτερα προδραστικοί. Εργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη, με τι ε, διαχειριστικέ αρχέ και βλέπουμε προβλήματα που είναι πέρα από τον ελεγχό μας όπως οι κρατικές ενισχύσεις και προσπαθούμε να καλέσουμε τους εμπειρογνώμονες και τις γάμα ΔΕΛΤΑ που είναι αρμόδιες στις συναντήσεις. Επίση ε, προσπαθούμε να στοχεύσουμε σε κάποια τέτοια ζητήματα όταν οι εθνικές αρχές δεν μπορούν να βασιστούν στα δικά τους εθνικά γραφεία. Και επίση ε, συνεργαζόμαστε πάρα πολύ με την Υπηρεσία Διευθυντικών Μεταρρυθμίσεων. Συνεργαστήκαμε πολύ μαζί τους, τους δώσαμε καθοδήγηση για το ποια project ε, θα πρέπει να τεθούν ω ε, προτεραιότητα και να ολοκληρωθούν από τη σκοπιά τη εφαρμογή και εργαζόμαστε και για το θέμα τη συμπληρωματικότητα. Δημιουργήθηκε το Ταμείο έύση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλα προγράμματα όπω ε, το Horizon ε, και έχουμε βάλει πάρα πολλέ δυνατότητε, αποφεύγοντα ε, τι επικαλύψεις για να έχουμε αυτά τα κοινά project έτσι λοιπόν νομίζω ότι είμαστε ιδιαίτερα προδραστικοί και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Όλες οι μονάδες μας, όλα τα τμήματά μας είναι κινητοποιημένα η απορρόφηση θα γίνει μόνο όταν μπορείτε να διασφαλίσετε ότι είναι ποιοτική. Αυτό είναι το μότο μας και γι' αυτό χρειάζεται συνήθως περισσότερο χρόνο από ό,τι θα θέλαμε. Όμως συμβαίνει, λαμβάνει η χώρα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες συστάσεις αναχώρας ε, και εκεί στοχεύουμε. Δεν μπορώ να μιλήσω για την μακροοικονομική ερωσιμότητα, είναι μια άλλη διαδικασία. Το πιο σημαντικό είναι να συνδεθούμε με τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη και να κάνουμε συγκεκριμένες επενδύσεις εκεί όπου χρειάζεται. Και επίση θα παρουσιάσουμε και μία έκθεση για τη συνοχή. Είχαμε το φόρουμ για τη συνοχή, πολύ ενδιαφέρον. Και εκεί θα δείτε τα συμπεράσματά μας ήδη για την περίοδο 2014-2020 και κάποιες ιδέες για το μέλλον ίσως. Που ίσως και να χρειαστεί να αλλάξουν. Όμω θα πρέπει να θυμόμαστε ότι πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Υπάρχουν πολλά καλά στοιχεία σε αυτή την περίοδο που θα πρέπει να συνεχιστούν ε, μετά το 2020. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι συνεννοούμαστε. Τέλος πάντων, ε, μάλλον δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα, αλλά κάποια στιγμή θα βρούμε την άκρη του νήματος. Mm. Ας περιμένουμε να δούμε τη μελέτη περιπτώσεων. Να δώσω τώρα το λόγο, γιατί περνάμε στη διαχείριση των κονδυλίων στις μελέτες περιπτώσεων. Λοιπόν, Πρέμπεν Γκρέγκερσεν από τη Δανία. Danish Business Authority. Πού είστε? Α, δεν σας έβλεπα. Παρακαλώ, καλώς ήρθατε και έχετε το λόγο. Does this work? Ε, είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. Έχω δουλέψει στα διορθωτικά ταμεία επί 20 χρόνια. Ποτέ δεν μου δόθηκε ευκαιρία να απευθυνθώ σε αυτή την επιτροπή. Χαίρομαι πάρα πολύ που με καλέσατε. Ευχαριστώ. Θα σας ε, περάσω ε, σε κάτι πάρα πολύ πεζό. Είμαι άνθρωπος που ασχολείται με τα πρακτικά που εφαρμόζεται, που εφαρμόζει τις, ε, τα προγράμματα. Ε, συμμετέχω και δηλαδή και στην διαδικασία της προετοιμασίας που πραγματοποιούμε. Επί της ουσίας όμως είμαι εγώ ένας από αυτούς που υλοποιούν και ως τέτοιος θα σας μιλήσω. Θέλω να σας πω ότι στη Δανία υπάρχει μία διαχειριστική αρχή που καλύπτει τα πάντα ε, σε σχέση με τα διαρθρωτικά ταμεία, δηλαδή το Ταμείο και, ε, Ανάπτυξης, το Κοινωνικό Ταμείο και το Ιντερεκ και αυτό οφείλεται στο μέγεθός μας, στο μέγεθος της χώρας μας. και τα ποσά που διαχειριζόμαστε επικεντρωνόμαστε στο πόσο σύνθετος είναι ο κανονισμός και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια κρίσιμη μάζα εμπειρογνωμοσύνης. Με δύο λόγια. Γνωρίζω ότι κατά πάσα πιθανότητα γνωρίζετε τη μορφή της ε, Δανίας. Οι κόκκινες κουκίδες είναι τα περιφερειακά κέντρα. Εκεί ε, Υπάρχουν τα, τα έξι μεγάλα κέντρα της χώρας. Σας το λέω αυτό γιατί ε, τα κέντρα αυτά και οι γραμματείες είναι βασικά στην κατανόηση του συστήματός μας. Εδώ ε, τα, οι χώροι ανάπτυξης ή τα βήματα ανάπτυξης, ε, τα κέντρα αυτά, είναι χώροι επιχειρηματικοί και εκεί ξεκινούν τα προγράμματα με ένα δοκιμαστικό φάκελο που τους έχει δοθεί για την επταετία. Δηλαδή γίνεται, αυτοί κάνουν την πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος, βλέπετε εδώ τα κόκκινα. Οι περιφερειακές γραμματείες προετοιμάζονται, προετοιμάζουν τις προσκλήσεις και τις προτάσεις για τα έργα. Αυτοί κάνουν τη δημιουργική δουλειά εκ μέρους της περιφερειάς τους. Κάνουν, οργανώνουν προσκλήσεις εντός του προγράμματος είτε πρόκειται για το κοινωνικό ταμείο, το ταμείο περιφερικής ανάπτυξης, ε, για κάποιο συγκεκριμένο τομέα έξυπνης εξειδίκευσης. Δηλαδή, με βάση την καινοτομία που χρειάζονται, ε, κάνουν την, ε, δική τους, το δικό τους σχεδιασμό, τη δική τους στρατηγική, εκτιμάζουν την πρόσκληση, ανακηρύσσεται ένας ή περισσότεροι νικητές και κατόπιν τα προωθούν τους, ε, αυτούς που επελέγησαν σε εμά τη διαχειριστική αρχή. Εμείς είμαστε αυτοί που κάνουμε τη σκληρή δουλειά, τη δύσκολη δουλειά. Εμείς είμαστε οι καημένοι, οι κακόμεροι, ενώ οι περιφέρειες κάνουν το ωραίο κομμάτι της δουλειάς, το δημιουργικό. Γι' αυτό τελικά στο διατάφτα πρέπει να πω ότι η οι ευφυείς επιλογές στο σύστημά μας στηρίζονται στο τόπο, ενώ το νομικό και το κομμάτι, το κομμάτι της παρακολούθησης ε, αφορά το γραφείο της ε, διαχειριστικής αρχής. Σημαντικό για την Επιτροπή σας πρέπει να είναι ότι όσον αφορά την υλοποίηση, σημασία έχει η ευθύνη, η λογοδοσία και η προόδος να έχουν ανατεθεί σε ανθρώπους που πρέπει να λαμβάνουν τις αποφάσεις. Είναι σημαντικό να υπάρχει πραγματική εταιρική σχέση, συνεργασία. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι εταίροι προκειμένου να λάβουν αποφάσεις και να ε, είναι υπόλογοι το, στην εφταετία της υλοποίησης. Εδώ υπάρχουν θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν ένα μάθημα, μια εμπειρία από την χώρα μου, την ταπεινή μου χώρα και ξέρω ότι τα μαθήματα που μπορώ να σας μεταφέρω από πλευρά σας ε, θα θεωρηθούν ότι προέρχονται από μια μικρή ε, χώρα που βρίσκεται στη βορειοανατολική περιοχή της Ευρώπης, αλλά ενδεχομένως κάποια από αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και διευρωπαϊκά. Αν δούμε τον ε, τομέα της απορρόφησης, αυτό είναι ένα σκέλος της, ε, του όλου εγχειρήματο. Γιατί η διαχειριστική αρχή πρέπει να ξέρει ότι αυτό που κάνει είναι αποτελεσματικό. Δηλαδή να μην ε, ε, ασχολείται μόνο με την απορρόφηση αλλά και με το αποτέλεσμα αυτής της απορρόφησης. Επίσης, ποιε είναι οι προσδοκίε των επενδυτών. Είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Εδώ υπάρχουν κίνδυνοι. Δεν μιλάμε για κάτι που δεν ενέχει κινδύνους. Αναλαμβάνονται κίνδυνοι. Υπάρχουν συγχρηματοδότε στην ε, Δανία οι οποίοι κινδυνεύουν τους, τα χρήματά του, όπω διακινδυνεύουμε και τα χρήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν κίνδυνοι εδώ. Μιλάμε λοιπόν για χαμηλό ποσοστό σφάλματος. Έχουμε την τύχη να το έχουμε επιτύχει αυτό για πολλά χρόνια. Η απορρόφηση είναι κομμάτι της καθημερινής δουλειάς, της υλοποίησης, της εξυπηρέτησης και της ε, ε, αντιστήχησης των ε, επιθυμιών των επενδυτών και αυτών οι οποίοι συμμετέχουν. Επίσης, ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν εγκρίνεται, είναι αυτό το οποίο θα δώσει το, αποτέλεσμα, το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει κανείς γιατί μερικές φορές έχεις, νιώθεις ικανοποιημένος για αυτό που κάνεις. Και λες ότι είναι πολύ εύκολο να πει κανείς ότι αυτό οφείλεται στην καλή διαχείριση των ποσών των ταμείων. Έχω προσπαθήσει να επιλέξω κάποια σημαντικά πράγματα. Πρώτον, η έγκαιρη έγκριση των προγραμμάτων και η έγκαιρη πρόσκληση. Δηλαδή, όταν θέλει κανείς να αρχίσει ένα πρόγραμμα στη Δανία, ξεκινάει το 2012 έτσι ώστε για να είναι πανέτοιμο να ξεκινήσει το 2014. Δεν ξεκινάς το 2014, δεν περιμένεις να έχει ολοκληρωθεί ο κανονισμός, να έχει διαβάσει τα πάντα. Πρέπει να ξεκινήσεις τον προγραμματισμό με ό,τι υπάρχει και κατόπιν, σύν το χρόνο, να προσαρμόζεσαι και να διορθώνεις και να είσαι έτοιμος για έγκριση όταν ξεκινάει η προγραμματική περίοδος. Στη Δανία τουλάχιστον ε, αυτό οδηγεί σε μια κατάσταση όπου η εταιρική σχέση του προγραμματισμού ξεκινά πριν καν γνωρίσουμε τους, τους κανόνες, πριν καν γνωρίσουμε αν υπάρχει προπολογισμό, πριν καν ξέρουμε αν, ε, πώς έχει οριστεί το ε, πεδίο πάνω στο οποίο θα κινηθούμε. Θα με ρωτήσετε ενδεχομένω. Τι λογική, ποια είναι η λογική του να υπάρχουν διαφορετικά ταμεία στη Δανία. Κοιτάξτε, η, τα, ταμεία, τα, η χρηματοδότηση αυτή στηρίζεται στον, στον τόπο. Υπάρχουν διάφορα κριτήρια του ΩΣΑ. Ένα από αυτά είναι πόσο ψηλή είναι η παραγωγικότητα, και εκεί βλέπει κανείς ότι έχουμε παραμεθόριες περιοχές και έχουμε περιοχές που είναι στην πρώτη γραμμή και περιοχές που, είναι, ε, που καθυστερούν. Πρέπει λοιπόν να δουλέψει κανείς επί τόπου για να μπορέσει να προωθήσει την ανάπτυξη στις ε, περιοχές που δεν είναι στο, στην πρώτη γραμμή. Αν υπήρχαν μόνο τέτοιες στην Ευρώπη θα δουλεύαμε εκ των, εκ των άνω προς τα κάτω. Αλλά αν πάμε σε περιοχές που είναι κάτω από τη Φραγκφούρτη, την Στοκχόλμη, την Κοπενχάγη, πρέπει να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το δυναμικό που χρειάζεται κάθε περιφέρεια. Κάθε περιφέρεια έχει δυνατότητα. Και επίσης πρέπει ευθύ εξ αρχής να είναι πλήρης η διοικητική βάση. Όταν το σύστημα είναι αποκεντρωμένο όπως είναι το δικό μας, θα πρέπει η περιφέρεια που θα αναπτύξει το έργο να ξέρει το πλαίσιο. Πρέπει να ξέρει ποια είναι τα κίνητρα που θα έχει και να ξεκινήσει. Και επίσης πρέπει να ξέρει ότι αν αργήσει θα υποστεί κάποια ποινή ή αν απομακρυνθεί από το πρόγραμμα. Υπάρχει δηλαδή, υπάρχουν εδώ μέτρα και σταθμά τα οποία ισχύουν, τα χρησιμοποιούμε για να παραμείνει στη σωστή πορεία το έργο. Επίσης, η απορρόφηση. Αν δεν είναι σωστή η απορρόφηση, αν καθυστερεί, θα τους το υπενθυμίσουμε στη Διαχειριστική Επιτροπή, όπου όλοι συμμετέχουμε και όπου συμμετέχουν οι πάντες. Ε, και εκεί πάλι ε, ε, εξετάζονται τα μέτρα και τα σταθμά. Το ίδιο ισχύει για τη συγχρηματοδότηση, για τους στόχους. Ε, πρέπει να υπάρχουν επαρκή κίνητρα, κατάλληλα εργαλεία ευθύ εξ αρχής. Κατόπιν είναι ο διάλογος. Για μένα είναι απλώς ένας διάλογος. Πολλά μπορεί να πει κανείς, πολλές όρους να χρησιμοποιήσει, αλλά ο διάλογος πρέπει να γίνει εκεί επιτόπου μεταξύ του, του, υπευθύνου, της Γενικής Διεύθυνσης Ρέτζου, της, της ε, ε, διαχειριστικής αρχής και ε, του υπευθύνου στο τοπικό επίπεδο και συμμετέχουν και οι ελεγκτές από το ευρωπαϊκό, το κρατικό και το τοπικό ελεγκτικό συνέδριο. Είναι μια διαδικασία που δεν σταματά, δεν μπορεί να είναι κάτι που γίνεται κάθε εξάμεινο, οποτεδήποτε θεωρήσουμε καλό να συγκαλέσουμε μια συνάντηση. Είναι κάτι που πρέπει να γίνεται διαρκώς, να διορθώνονται τα σφάλματα. Εγώ από πλευράς μου μπορώ να πω ότι αφού δουλεύω σε αυτό το χώρο από το 94, 20 χρόνια, ότι ο διάλογος που είχαμε με τους υπευθύνου της Κομισιόν, με το ελεγκτικό συνέδριο, με τους ε, ελεγκτές που είναι υπεύθυνοι επιτόπου, ε, ήταν πάντοτε εξαιρετικός, δηλαδή πάντοτε είχε στόχο να είναι αποτελεσματικός εκεί, στο πεδίο. Και αυτό ήταν κρίσιμη σημασία για κάποιες από τις επιτυχίες που γνωρίσαμε. Τώρα, επανέρχομαι στην απορρόφηση για να εξασφαλίσω ότι θα τη συζητήσουμε την απορρόφηση. Ήδη σας είπα ότι όταν είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινά το πρόγραμμα εγκαίρως. Είναι σημαντικό για μένα να ξέρω ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα που ε, επικεντρώνεται σε κάποιες σημαντικές προτεραιότητες. Καινοτομία, επιχειρηματικότητα, ε, η δημιουργία δυνατοτήτων στο κοινωνικό ταμείο, μακροχρόνιες, βραχυπρόθεσμες κτλ. Αλλά το καλύτερο που μπορεί κανείς να κάνει όσον αφορά την απορρόφηση είναι να σχεδιάσει προγράμματα που καθοδηγούνται από τη μακροχρόνια ανάπτυξη. Δηλαδή, όσο ε, λιγότερες είναι οι κρίσεις και οι οξύτητες στη μακροχρόνια υλοποίηση, τόσο το καλύτερο. Ήτι, e το πρόγραμμα πρέπει να καθοδηγείται από μια ευρεία συνεργασία, μια ευρεία εταιρική σχέση, όπου όλα τα μέρη να έχουν τον ίδιο στόχο σε επίπεδο πολιτικό, σε επίπεδο οργανωτικό και σε επίπεδο υλοποίησης. Όλοι πρέπει να συμφωνούμε ότι μα ενδιαφέρει η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα ή όποιος, όποιος στόχος έχουμε θέσει. ώστε το πρόγραμμα να υλοποιηθεί με, μια, με ένα μακροπρόθεσμο, με μια μακροπρόθεσμη προοπτική. Επίσης, οι περιφέρειες αν ε, ε, παρακολύουν το πρόγραμμα πρέπει να ανακληθούν στην τάξη. Δηλαδή πρέπει να κινηθούν γρήγορα μέσω των προσκλήσεων και τα λοιπά, να μπορούν να αντιδράσουν απέναντι στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Υπάρχει ένα σύστημα τριμηνιαίο που έχουμε ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της πρόοδου με τις γραμματείες. Είναι ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να προσέξετε. Όταν βλέπετε ε, ε πρώιμα νούμερα για τα κονδύλια υποχρεώσεων στα κράτη-μέλη, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι δαπάνες ενεργές, μπορεί να είναι παθητικές. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε από ένα κράτος μέλο, για να δούμε αν πηγαίνει καλά ένα πρόγραμμα, πόσε συμβάσεις έχουν συναυθεί. Γιατί με τα χρόνια παρατήρησα ότι εγώ θεωρούμε ότι καθυστερώ την αρχή της προγραμματικής περίοδου γιατί μετρώνται μόνο οι συμβάσεις και καμιά φορά συγκρινόμουν με κράτη-μέλη τα οποία κρατούσαν, ε, μετρούσαν τις δεσμεύσεις τους και μου λέγανε «Α, καθυστερείς, καθυστερείς, τι συμβαίνει». Αυτή είναι μια σημαντική διάκριση. Αν μιλάμε σαφώς για την απορρόφηση, και αυτό είναι το θέμα μας τώρα, θα πρέπει να μιλάμε για τα, τον αριθμό των συμβολέων, των συμβάσεων που έχει υπογράψει η διαχειριστική αρχή. Διότι εκεί μπορεί να μετρηθεί η προόδος. Αν απλώς μιλάει κανείς για γενικές δεσμεύσεις, αυτά όλα μπορεί να είναι παθητικά και να παραμείνουν έτσι για μεγάλο διάστημα. Να είναι και αντιπαραγωγικά στη χειρότερη περίπτωση. Πρέπει επίσης όλο και περισσότερο να έχει κάνει κανείς διάλογο για κάθε μία προτεραιότητα με τις περιφέρειες ή με όποιον είναι αρμόδιος να ε, ζητά πρόσκληση από πολύ ενδιαφέροντος. Και έχουμε τέτοιες επαφές κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα. Πριν κλείσω αυτό το μέρος, θέλω να πω το εξής. Υπάρχουν μέρες που αισθάνομαι ότι η, η βασική μας γλώσσα έχει, μας έχει ξεπεράσει. Πάω εγώ στη, γλώσσα, στη χώρα, στην πόλη μου ή σε άλλες πόλεις και ακούω την ευελιξία, την απλούστευση. Είναι γενικοί όροι που όλοι, όλοι συμφωνούμε, αλλά κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς σημαίνουν. Όλοι λοιπόν είμαστε εκεί, ακούμε, κουνάμε το κεφάλι μας καταφατικά, συμφωνούμε σε πράγματα που όλοι θεωρούμε ότι είναι θετικά. Ε, ε, εκ των άνω, εκ των κάτω, ευελιξία, προσέγγιση, απλούστευση, όλα αυτά μπορούμε να τα πούμε. Και μπορούμε να παίζουμε μπίνγκο στην ουσία πρέπει να γνωρίζει κανείς και θα σας δώσω και συγκεκριμένο παράδειγμα ότι κάθε ένα από αυτά τα πράγματα πρέπει να έχουν ένα νόημα στο πεδίο ώστε και εγώ και ο υπουργό μου να γνωρίζουμε τι σημαίνει ευελιξία. Για κάποιους ευελιξία σημαίνει ότι η διαχειριστική αρχή κάθε τόσο μπορεί και να μην δουλεύει και να περνάει καλά. Ναι, και αυτό το, το νόημα μπορεί να έχει η λέξη ευελιξία, αλλά υπάρχει και μια δύσκολη μορφή ευελιξία. Για μένα ευελιξία μπορεί να είναι ότι θα δεχτώ την άποψη του κυρίου Πόπεν για να ε, μου δώσει έγκαιρη έγκριση. Α πούμε, δεν μου άρεσε το αστικό ζήτημα. Εμάς στην Δανία δεν, δεν μας άρεσε πολύ αυτό το αστικό σύστημα γιατί εμεί τα είχαμε αυτά λύσει πριν τα καν τα σκεφτεί η Κομισιόν. Θα, είπαμε ότι ε, δεν μας χρειάζονται αυτά άσε 5% στην άκρη για το αστικό. Αλλά έλεγε ο κανονισμό, το προέβλεπε αυτό. Θα μπορούσα επί δύο χρόνια να το συζητώ αν το χρειάζομαι, το χρειάζομαι και τελικά ποτέ δεν θα μου ενέκριναν το πρόγραμμα. Αλλά αποφάσισα να δείξω ευελιξία και να πω ναι θα βάλουμε το 5% για να σα ικανοποιήσω και εσά και την Κομισιόν και μετά θα το υλοποιήσουμε. Και μετά είχαμε την πρώτη έγκριση, πρώτη από οποιοδήποτε άλλο κράτο μέλος. Αν είχα επιμείνει ότι δεν μου αρέσει αυτό το αστικό, θα περίμενα επί χρόνια. Αυτό είναι μια άλλη ευελιξία. Ευελικτός απέναντι στο ευρωπαϊκό σύστημα για να μπορώ να πετύχω την έγκαιρη έγκριση. Χαίρο, ε, λυπάμαι που αναφέρω το όνομά σας κύριε Πόπενς, αλλά ένας καλός τρόπος συνεργασίας είναι να δείξει κανείς ευελιξία κατά την υλοποίηση για να κάνει τα πράγματα εγκαίρως. Δεν αν είσαι διαχειριστής διαρθρωτικών ταμείων, όσο πιο ανυπόμονος είσαι, ακόμα και κακός να είσαι, όσο ε, αν εργάζεσαι με ανυπομονησία είναι καλό. Θα σας, όλοι μπορείτε να διαβάσετε τις διαφάνειές μου, θα φτάσω στο τελευταίο στοιχείο. Αυτό σημαίνει η κατεύθυνση προς το ε, αποτέλεσμα, η επικέντρωση στο αποτέλεσμα. Σας έλεγα γενικές, γενικές, γενικές όρες το αποτέλεσμα δεν είναι πολύ σεξι λέξη. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει κανείς να ανταποκριθεί σε ένα πρότυπο που κάθε είσοδος χρήματος πρέπει να σχετίζεται με μια κρίσιμη δραστηριότητα, με ένα, αποτελέσματα, με ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αυτό θα πει αποτέλεσμα επιτόπου. Αντί λοιπόν να μιλάμε όλη την ημέρα στις Βρυξέλλες ή στην Κοπενχάγη για το τι σημαίνει καθοδηγούμε από το αποτέλεσμα, στο γραφείο μου αυτό σημαίνει όταν συζητώ με τα έργα. Τα δικά μου έργα στο όνομα αυτού που όλοι συμφωνούμε, στο όνομα του αποτελέσματος, πρέπει να πετύχουν τις κρίσιμες, τα κρίσιμα, τους κρίσιμους δείκτες. Παλιά λέγαμε δώσουμε 500 εκατομμύρια θα κάνω ένα θαύμα. Όχι, τώρα έχουμε βήματα στην πορεία. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί αν πάμε προς τα πίσω, βλέπετε ότι τώρα έχω καλύτερο αποτέλεσμα. Ενδεχομένως όμως για κάποιο διάστημα ίσως να πληρώσω λίγο στον τομέα της απορρόφησης γιατί κάποιος μαθαίνει ένα μάθημα. Περιμένω μέχρι να μάθει το μάθημα, μετά θα το τιμωρήσω και θα προχωρήσω στον τομέα της απορρόφησης. Ενώ τώρα πάει, το, όλη η προσοχή στρέφεται στο μέγιστο αποτέλεσμα. Και ο απλός δημόσιος υπάλληλος, και ένα μικρό κράτος μέλος, μιας διαχειριστικής αρχής έτσι εργάζεται καθημερινά. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες που έχουμε, να τους ευχαριστήσω θερμότητα για τη συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια. Δεν λέω ότι διασκεδάσαμε, αλλά ήταν μια ενδιαφέρουσα συναλλαγή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκρέγκες. Χαιρόμαστε και εμείς που είστε εδώ. Κυρία Γκρό. Α, ποιος θέλει το λόγο. Κύριε Σαββά, ευχαριστώ. Συγγνώμη που διέκοψα. Επειδή θα φύγω, δεν μπορώ να περιμένω να θέσω τις ερωτήσεις μου στο τέλος. Ε, ωραία, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο τώρα. Δεν έχω ε, κάποιες επικρίσεις να εκφράσω, αλλά να κατάλαβα καλά. Είπατε είστε εδώ για πρώτη φορά. Ευτυχώς που ήρθατε και πολύ αργήσατε. Και ο λόγος που το λέω είναι γιατί Έτσι ακριβώς θα έπρεπε να αξιοποιούνται τα χρήματα που δίνουν. Και έχω και μία ερώτηση, γιατί είπατε ότι πρέπει να γίνεται διάλογος με τις περιφέρειες συνεχώς, με τους ανθρώπους επιτόπου. Αυτό περιλαμβάνει και αμφίδρομη επικοινωνία, σε σχέση με τις βασικές αρχές δηλαδή. Τους όρους τους γνωρίζουμε όλοι. Τι καταλαβαίνουμε όμως όταν ακούμε όρους ε, όπως ευελιξία ή κάτι άλλο τέλο πάντων. Έρχεστε, όχι καθημερινά, αλλά τέλο πάντων ε, σε, κάθε, σε τακτά διαστήματα, 72 άλλος. Για να καταλάβουν ε, οι συνομικτές σας τι θα πει καλύτερες επιδόσεις. Ναι και η συνάδελφος Αγιάλα είχε μια ερώτηση. Ναι, ευχαριστώ. Δεν είναι πρώτη φορά. Εσείς ναι. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχής γιατί μας παρουσιάσατε την εμπειρία ενός υπαλλήλου. Αν θέλετε που έχετε αντιμετώπιση με την πολυπλοκότητα. 94, άρα μπορείτε να μας μιλήσετε για, γιατί ξέρετε πολύ, πολλούς κύκλους, ε, πώς πήγε μέχρι τώρα η διαδικασία από το χειρότερο στο καλύτερο ή ανάποδο. Σπαθείτε να λύσετε τα προβλήματα. Έχουμε μιλήσει με εκπροσώπους της Δανέσκης Κυβέρνησης. Προσπαθώντας να έχουμε ακριβώς ε, το result oriented budgeting. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι με ποιους δείκτες καταφέρνετε να έχετε αυτά τα βραχυπρόθεσμα αποτελεσματα short term results, δηλαδή τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα καθημερινά και πώς αυτό το συσχετίζεται με τα, με τα μακροχρόνια αποτελέσματα, long term results. Γιατί αν μιλήσουμε τους εκπρόσωπους της ε, δανέσκης κυβέρνησης και κάποια στιγμή το κάναμε αυτό, μας είπαν ότι δεν έχουν λύσει τα προβλήματα, το αντίθετο. Εντάξει, μπορεί να μην είναι συγκρίσιμα τα θέματα. Εμεί έχουμε 40 εκατομμύρια από υπέρ Αλλά τέλο πάντων, να δούμε ποιε είναι οι καλέ πρακτικέ. Uh, yes. Ευχαριστώ. Ναι. Να ξεκινήσω με το περιφερειακό στοιχείο. πάντα υπάρχει μια γραμματεία που υποστηρίζει και η οποία απαρτίζεται από πολύ ικανούς ε, ανθρώπους. Και από την αρχή συμμετέχουν ε, όταν καταρτίζονται τα προγράμματα. Σε ό,τι αφορά τους κανόνες επιλεξιμότητας και όλους τους άλλους κανόνες πρέπει να τα ξέρουν το ίδιο καλά όσο και η διαχειριστική αρχή σχεδόν. Γιατί αλλιώς οι συμβουλές που δίνουν στους διαγωνισμούς, δηλαδή όταν κάνουν διαγωνισμούς, θα έλειπαν στοιχεία. Άρα έρχονται σε επαφή τακτικά μαζί μας ε, όταν κάνουν διαγωνισμούς για τεχνικά ζητήματα. Το προσωπικό που έχω εγώ στο επίπεδο ΜΕ και αυτό που υπάρχει σε επίπεδο γραμματιακό συνεργάζονται πολύ καλά. Το θέμα είναι αν υπάρχει ένα δύσκολο ζήτημα, αν υπάρχουν πολύ κανόνες κρατικών ενισχύσεων, έρχονται σε εμά και ζητούν ε, γνωμοδότηση, την άποψή μας, νωρίς, σε πρώιμο στάδιο, για να μπορέσουν να καταθέσουν κάτι το οποίο θα είναι θεμητό. Άρα έχουμε αυτή την τακτή επικοινωνία, τακτική επικοινωνία. Επίσης, Υπάρχουν εκπρόσωποι σε αυτά τα φόρου. έχουμε εκπροσώπους από χώρους γνώσης. Συνολικά έχουμε 21 μέλη. Όλοι αυτοί έχουν μελετήσει το θέμα, του αν αυτή η έξυπνη εξειδίκευση προχωρεί σωστά είναι εντάξει. Αυτό συμβαίνει διαρκώς. Δεν υπάρχει τρόπος αυτό να διεκπαιρεωθεί μέσα σε δύο ώρες. Το άλλο θέμα. Έχετε δίκιο. Μπορεί να είναι δύσκολο. Κάνουμε όμως στη Δανία δύο πράγματα όσον αφορά τα αποτελέσματα. Για το χρόνο μετά το αποτέλεσμα. Ας πούμε το κοινωνικό ταμείο ή ένα καινοτόμο έργο. Καθορίζουμε τους δείκτες απόδοσης ανάλογα με το πρόγραμμα και ανάλογα με τα κριτήρια με τα οποία δουλεύουμε. Αν ένα έργο λοιπόν δεν καλύπτει τα κριτήρια. Ας πούμε ένα κριτήριο καινοτομία είναι ότι θέλουμε στη Δανία να υπάρχουν περισσότερες καινοτόμες επιχειρήσεις αν αυτός δεν είναι στόχος του προγράμματος, τότε είναι παραπλανητικό αυτό και το λέμε. Ας πούμε ότι το βραχυπρόθεσμα, το αποτέλεσμα θα είναι ότι περισσότερες επιχειρήσεις θα αναφέρουν ότι αισθάνονται πιο καινοτόμες. Εμείς όμως στηριζόμαστε στους αριθμούς εγγραφής κατά αυτών που συμμετέχουν. Δηλαδή τους περνάμε από τη στατιστική υπηρεσία και μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις εταιρείες που συμμετείχαν στο έργο και να τις συγκρίνουμε με άλλες εταιρείες που δεν συμμετείχαν. Δηλαδή βλέπουμε ε, ποιο είναι το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν κάνουμε απευθείας χορηγίες σε εταιρείε. Εμείς λειτουργούμε σε πλαίσια συστημάτων. Παρακολουθούμε όμως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες για να δούμε πώς προσλαμβάνουν σε σχέση με αυτούς που δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα και έχουμε θετικά αποτελέσματα και μακροπρόθεσμα στην περίοδο 7-13 σε σχέση με μια ομάδα ελέγχου μη συμμετεχόντων τη Να ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι τιμή μου να είμαι εδώ σήμερα. Λυπάμαι που δεν είχα ε, μια καταλεκτική ημερομηνία για να παρουσιάσω το έγγραφο που είχα προετοιμάσει και δεν βρίσκω τις διαφανίες μου στη έγγραφα που έχουν διανεμηθεί, αλλά καθώς ε, τώρα τα έχετε εσείς στη διάθεσή σας, ε, θα σας ε, ζητούσα να τα μοιράσετε αυτά τα slides. Πριν να ξεκινήσω, θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποιες ιδέες που μου ήρθαν από τους προλαλήσαντες κυρίως σε ό,τι αφορά το ελεγκτικό συνέδριο, δηλαδή να επικεντρωθούμε στη λογική της παρέμβασης και οι έλεγχοι που γίνονται να μην χάνουν ποτέ από το νου τους ότι αυτά τα κονδύλια θα πρέπει να βλέπουμε ποια είναι τα αποτελέσματα που αφήνουν τόπου. Είναι ε, η πολιτική που είχε ακολουθήσει μακροπρόθεσμα και ε, η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη και οι εταίροι τους. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στη λογική της παρέμβασης, στη στρατηγική της παρέμβασης και στα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε. Θα ξεκινούσα τώρα με μια πρώτη διαφάνεια. Ευχαριστώ τον δανό συνάδελφο γιατί πράγματι μας ε, έδειξε ε, πόσο αποτελεσματική είναι η οργάνωση και εγώ προερχόμενη από μια χώρα που είναι διερεμένη στα δύο μπορώ να σας πω ότι στις πιο αναπτυγμένες χώρες έχουμε ε, λιγότερους σπόρους αλλά υπάρχουν πολλές ε, ικανότητες για το παραγωγικό σύστημα. Σίγουρα η απορρόφηση και η ικανότητα παραγωγής αποτελεσμάτων είναι μεγαλύτερη. Η Ιταλία όπως ξέρετε έχει όλες τις περιφέρειες ε, του Βορρά σε μια πλεονεκτική θέση, ενώ οι περιοχές του Νότου, οι περιφέρειες του Νότου που επιφελούνται περισσότερο από τα κονδύλια είναι αυτές που συνάντησαν μεγαλύτερες δυσκολίες. Έτσι λοιπόν έχουμε μια διτή εμπειρία και έχουμε μια διτή εμπειρία επομένως για το πώς οι διαχειριστικές αρχές μπορούν να βοηθήσουν τους δικαιούχου. Βλέπουμε εδώ πως πήγε περίοδος 2007-2013 για μας, μια περίοδο αρκετά δύσκολη, η κρίση ε, ουσιαστικά χτύπησε πολύ σκληρά την Ευρώπη, τα διαρθρωτικά ταμεία και το είπε αυτό και έκθεση της Κομισιόν, χρησιμοποιήθηκαν και για να αντιμετωπιστεί η κρίση αυτή έτσι λοιπόν με κάποιο τρόπο έχασαν τον πρόσθετο χαρακτήρα τους. Παρόλα αυτά η Ιταλία κατόρθωσε να έχει πλήρη απορρόφηση και αυτά είναι τα οικονομικά στοιχεία. Βλέπουμε το 2014 είμαστε ανάπτυξη 70%, το 2015 στο 80,5%, 2016 στο 98,1% και το 2017 το σημείο του κλεισίματος φτάσαμε στο 101%. Αλλά αν ε, θεωρήσουμε και τις αναστολές ε, φτάσαμε ε, σε ένα 4% απορρόφηση. Το θεωρούμε ότι είναι καλό το αποτέλεσμα γιατί είναι το μεταξύ. Έχουμε ε, διαφορετικέ μεταρρυθμίσει. προωθήσαμε το περιβαλλοντικό κεκτημένο, προσαρμόσαμε τα για συμβάσει συμβάσεις και έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και ενισχύσαμε όλα τα συστήματα ελέγχου του κράτου μα. Ακριβώ τώρα, επειδή δεν θέλω να μιλήσω για οικονομική απορρόφηση, θέλω να σας δείξω και ένα γράφημα ε, για τις δαπάνες, γιατί ποτέ δεν ξεχάσαμε τους θεματικούς ε, στόχους και αυτή είναι η λογική της παρέμβασης, ε, δηλαδή από τα 30,4 εκατομμύρια του στόχου της σύγκλησης βλέπετε εδώ έχουμε τους κύριους τομείς Λοιπόν, από αυτά 30,4 δις, οι τομείς που προώθησαν ε, ήταν ε, η καινοτομία, η εκπαίδευση, το περιβάλλον, η πρόληψη του κινδύνου, ο τουρισμός με 5,6 ε, για την έρευνα, 4,2 για το περιβάλλον και την πρόληψη κινδύνου, ε, συγγνώμη, για την εκπαίδευση μάλλον ήταν αυτό το ποσό. Θα έλεγα λοιπόν ότι όπως είπε και ο Δανός συνάδελφος, σε τι χρησιμεύει αυτή η πολιτική, γιατί υπάρχουν αυτά τα πολιτικά και αστυνομικές περιοχές, γιατί είναι μία ε, πολιτική περιφερειακή η οποία αντιμετωπίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες ανάπτυξης της περιφέρειας. Εγώ λοιπόν επικεντρώθηκα ιδιαίτερα γιατί σε αυτό μου φαινόταν ε, ότι είναι το κύριο θέμα που πρέπει να δούμε. Επικεντρώθηκα λοιπόν στις προβληματικές που κατά κάποιο τρόπο ε, δημιούργησαν ε, τα προβλήματα στην απορρόφηση. Ανέφερα ήδη κάτι που ήταν η οικονομική κρίση. Στην οικονομική κρίση θα ήθελα να συμπεριλάβω και το γεγονός ότι ταυτόχρονα είτε η Ιταλία είτε άλλες χώρες ε, βίωσαν όλες τις πολιτικές ε, του ε, fiscal compact. Δηλαδή ουσιαστικά είναι δύσκολο να σεβαστείς τις απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας ακόμη και για την τοπική αυτοδιοίκηση, τους φορείς της οπτικής αυτοδιοίκησης ήταν δύσκολο όλα αυτά. Ήταν δύσκολο όλο αυτό υπέφεραν πάρα πολύ από αυτό το στραβισμό, αν θέλετε να το πω έτσι. Δηλαδή, από την άλλη πρέπει να κάνεις κάποιες δαπάνες και από την άλλη πρέπει τελικά ε, να σεβαστείς πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες για την εξυγένση του προϋπολογισμού. Αυτό συνεισφέρε ε, σε αυτό συνεισφέρει και δύο ο μηχανισμό των διαφορετικών ταμείων. Ο μηχανισμό ε, τη επιστροφή. Δηλαδή, ε, δεν είναι, υπάρχουν κάποια κονδύλια που ο άλλος τα κρατά κατά μέρους. Ε, έτσι λοιπόν, όταν είχαμε την ημοκρομική κρίση δεν ήταν ε, τόσο ισχυρός αυτός ο σπονδύλος γιατί έπρεπε ουσιαστικά να επιστραφούν αυτά τα κονδύλια. Βέβαια το ότι φτάσαμε εμεί στο 100% σημαίνει ότι έχει απορροφήσει τα πάντα. Ίσως όχι ε, μέσα στο χρόνο με τον οποίο έπρεπε, όμω αυτό είναι ένα θέμα που έχει αντίκτυπο στον κοινωνικό προπολογισμό. Όλο πρέπει να έχουμε κατά νου ότι όλοι μαζί είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ μεγάλη κρίση. Και έτσι λοιπόν αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου όταν ε, αναλύουμε τα δεδομένα αυτά. Μια άλλη δυσκολία που τη βλέπετε σε, αυτό το, σε αυτή τη διαφάνεια ήταν ε, ε, οι προθεσμίες και οι κανονισμοί. Ε, αναγνωρίζω ότι στα κράτη-μέλη, ε, ούτε τα κράτη-μέλη του Κομισιόν το 2007-2013 μπορούσαν να κάνουν μια εγκαιρή διάγνωση των δυσκολιών. Θα πω όμως ότι εδώ βλέπετε πολύ καλά πως όταν η Ευρώπη από το 1994 μέχρι σήμερα επένδυε στις πολιτικές συνοχές, πώς ήταν οι κανόνες το 1994 και πώς αυξήθηκαν οι κανόνες στο 2007-2013. Ε, δηλαδή, όπως έλεγε ο συνάδελφος, αντί να έχουμε απλούστευση, τι, σε τι φτάσαμε, στο να έχουμε 5.000 σελίδες κατευθυντηρίων γραμμών και αποσαφηνήσεων αυτό φυσικά έχει αντίκτυπο. Αν σκεφτούμε στη συνέχεια ότι πολλέ από τι χώρε μα έχουν μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει, που είναι οι κύριοι δικαιούχοι των διαφορετικών ταμείων, για τι ΜΜΕ ένα τόσο πολύπλοκο σύστημα σίγουρα δεν ευνοεί. Δεν ευνοεί την ταχεία απορρόφηση. Τα μέτρα τώρα που προσπάθησε να πάρει η Ιταλία για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της περίοδου 2007-2013 που εμφανίστηκαν ξεκάθαρα από το 2011 και μετά, ίσως με κάποια δευτέρηση όπως σας είπα, είναι αυτά που ε, είδαμε στις ειδικέ συστάσεις αναχώρα. χώρα. Ε, σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε πως από το 2011 μέχρι το 2014 είχαμε συγκεκριμένες συστάσεις. Το 2016 υπόθηκε ότι φτάνουν τα μέτρα που έχουν ε, ληφθεί, όμως ε, απλώς ε, ουσιαστικά έπρεπε να κλείσουμε εκείνες τις διαδικασίες μεταρρύθμισης που είχαμε ξεκινήσει για την πολιτική συνοχής. Τώρα, για να το ξαναδούμε νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε το εξή. Σε μια χώρα που είναι η δεύτερη χώρα παραλήπτης της πολιτικής συνοχής που έπρεπε να διαχειριστεί 46 δι σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης και κάποιες από τις ε, πιο πολυπληθείς ε, περιφέρειες αν και είναι πολύ οικονομικές ε, ενεργά, αλλά είναι δύσκολη η διαχείρισή τους, κατέληξαν να έχουν πλήρη απορρόφηση. Και Ήδη σα τι ε, ανέφερα, έχουμε τα προβλήματα που ήταν η κρίση, ο μηχανισμός της επιστροφής κατόπιν ένα χαμηλό επίπεδο ολοκλήρωσης ε, της διακυβέρνησης σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό γιατί πολλοί έλεγχοι επικαλύπτονταν και όντως επιβαρύνουν την ε, διαχείριση. Ένα τελευταίο σημείο που δεν ανέφερα, συγγνώμη πάω προς τα πίσω, είναι ότι σε κάθε περίπτωση υπήρχε και ανικανότητα από την πλευρά της διοίκησης, ε, δηλαδή δεν επαρκούσε η ικανότητα της διοίκησης. Και στην ε, Συμφωνία Εταιρική Σχέσης που εγκρίθηκε καθυστερημένα, αναφέρθηκε και αυτό το θέμα από το ελεγκτικό συνέδριο για την περίοδο 2014-2027. Μειωμένη λοιπόν διοικητική ικανότητα είχε ε, πάρα πολύ μεγάλες συνέπειες. Ελήφθησαν ε, βέβαια πάρα πολλά μέτρα για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη αυτή. Ποια είναι τα μέτρα που πήραμε. Καταρχήν, την ε, μείωση της εθνικής χρηματοδότησης. Καταρχήν μιλούσαμε για εθνική χρηματοδότηση. Τώρα, τι σημαίνει, ε, ουσιαστικά δεν μιλάμε για, δεν προβλέπεται ε, αυτή η πολιτική από όλε τις προγράμματα χρηματοδότησης της Κομισιόν, όμως η Ιταλία πάντοτε σε χρηματοδοτούσε αυτό το έκανε ενεργοποιώντας ένα σχέδιο δράσης για τη συνοχή. Ε, δηλαδή, ε, έπρεπε να έχουμε προγράμματα επενδυτικά τα οποία αναφέρονταν στην πολιτική συνοχής και έδιναν στις περιφέρειες την ευκαιρία όλη η συγχρηματοδότηση που στην αρχή είχαμε δεσμευτεί να δώσουμε στην Κομισιόν να μπορεί να παρακολουθεί το πώς δαπανώνται αυτοί οι πόροι που ήταν εθνικοί πόροι και έτσι τιμήσαμε τη δέσμευση που είχαμε αναλάβει για την συγχρηματοδότηση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα μέρος αυτών ε, των κονδυλίων ε, δημιούργησαν και ένα αντισταθμιστικό ταμείο, ένα ταμείο αποζημίωσης ε, που ουσιαστικά προσπαθούσε να βοηθήσει κάποιες περιφέρειες που αντιμετώπισαν δυσκολίε λόγω του Συμφώνου Σταθερότητα. Επίση, όνομα με τι περιφέρειε κάναμε αυτό το διάλογο, ε, ένα συνεχή καθημερινό διάλογο, στον οποίο αναφέρθηκε και η Δανία. Εκεί συμμετέχουμε ισότιμα για να καλύψουμε το χαμένο χρόνο και δρόμο και με τη συμμετοχή της Κομισιόν και με συγκεκριμένη tax force για τα προγράμματα που είχαν καθυστερήσει περισσότερο για τη Σικελία, την Καμπανία και την Καλάμπρια. Και ε, κάτι άλλο που είναι επίσης ε, σημαντικό είναι η ενίσχυση του ρόλου της ελεγκτικής αρχής ε, ακριβώς για να έχουμε πιο εύρωστους ελέγχους ε, στο κράτο μέλος και για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε στους ελέγχους των Κομισιόν ένα πολύ χαμηλό ποσοστό λάθους και ε, αυτό ακόμη και αν περάσαμε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες με την αναστολή των ε, πληρωμών. Χρειαστήκαμε από 16 έως 36 μήνες ε, για τους ελέγχους αυτούς και φυσικά δημιουργήθηκαν τεράστιες δυσκολίες. Πρόκειτο για ελέγχους που ποτέ τελικά δεν σκόπευαν στο να παρουσιάσουν ένα αποτέλεσμα, αλλά είχαν να κάνουν με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με όλους αυτούς τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές και με προσανατολισμούς που για τους ελεγκτές, ε, είτε τους εθνικούς είτε τους ελεγκτές κομισιών, είναι νέα ε, στοιχεία απαιτήσεων και φυσικά προσθέτουν μεγαλύτερες δυσκολίες, κάνουν πιο δύσκολο το έργο της ε, διαχειριστικής αρχής. Ουσιαστικά ήταν έγινε η συνάντηση των διευθυντών νομίζω ότι υπόθηκε αυτό το ζήτημα. Στη συνέχεια προσδιορίσαμε ε, τι σημαίνει θεσμική διακυβέρνηση. Δημιουργήσαμε έναν οργανισμό, τον οποίο σας ανέφερα, και διαχωρίσαμε τον προγραμματισμό από την υλοποίηση. Δημιουργήσαμε ένα φορέα που να μπορεί να παρακολουθεί βήμα-βήμα την εφαρμογή. Επίσης προσλάβαμε 120 άτομα ε, ειδικού ε, για τα διαρθρωτικά τομεία για να βοηθήσουν ε, τη δίκηση ε, στο συντονισμό και για να βοηθήσουν τις διαχειριστικές αρχές. Ε, ε, είχαμε 29 σχέδια διοικητικής ενίσχυσης. Έτσι λοιπόν, κάθε κεντρική διοίκηση είχε ένα τέτοιο σχέδιο διοικητικής ενίσχυσης και εδώ βασιστήκαμε πάρα πολύ στο θέμα της διαφάνειας. Το Open Cohesion, νομίζω το ξέρετε όλοι, έχει βραβευτεί στην Ευρώπη, διαφάνεια, διάθεση πληροφοριών και η δυνατότητα να ε, μπορέσουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν και σε αυτή την ευρωπαϊκή πολιτική και το τι μπορεί να, ενημερωθούν για το τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη. Ε, γιατί μπήκαμε και μέσα στα σχολεία με το πρόγραμμα αυτό. Επίσης, ε, δεν αναφερθήκαμε μόνο στο θέμα της χρηματοδότησης, αλλά και στα αποτελέσματα που φέρνουν αυτές οι πολιτικές στις περιφέρειες. Αποτελέσματα που σας παρουσίασα σήμερα. Τώρα, ίσως ε, να ξαναγυρίσω πίσω. Θα ήθελα να αναφερθώ στα σχέδια ενίσχυσης της δίκησης. Αυτό είναι ένα εργαλείο που μόνο η Ιταλία έχει στην Ευρώπη και γίνεται ο συντονισμός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δηλαδή έχουμε πολύ υψηλό επίπεδο συντονισμού συμμετέχουν ε, και οι περιφέρειες ε, σε αυτό και η κάθε περιφέρεια έπρεπε να κάνει μια αξιολόγηση για τις δικές της ανάγκες και για τη διοικητική της ικανότητα. Έπρεπε να συντάξει ένα σχέδιο για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα όχι μόνο στη διαχείριση των πόρων, αλλά και σε όλα τα συναφή με τη διαχείριση των πόρων. Όπως ε, είδαμε, χρειάζονταν πολλά να γίνουν επειδή ήταν πολύπλοκο όλα αυτά. Και για την περίοδο 14-2020 ήθελα να πω το εξής. Εμείς ε, έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη γλώσσα όταν μιλάμε για τα διαρθρωτικά ταμεία. Συμμετείχαμε με πολύ μεγάλη προσοχή στις εργασίες της ομάδας υψηλού επίπεδο για την απλούστευση και στις εργασίες του Όμνιμπου. Όμως θεωρούμε ότι σε επίπεδο απλούστευσης ε, και είδατε το γράφημα που σας έδειξα πριν, δεν έχουμε καταλήξει σε καλά αποτελέσματα. Σας ε, το επισημαίνω εκ νέου, γιατί πρέπει να το έχουμε κατά Πρέπει να εργαστούμε πάρα πολύ σε αυτό το θέμα της απλούστευσης, γιατί όταν ε, η Κομισιόν ε, ουσιαστικά ζητά να γίνουν επενδύσεις από τα κράτη-μέλη, κοιτάξτε, θα πρέπει ε, να δει και το εξή, γιατί η έχει αυτή την ανησυχία μεταξύ των πρωτοτήτων, ότι θα πρέπει πάντοτε να σκέφτεται πώς θα διευκολύνει λίγο τη ζωή των άμεσων δικαιούχων και πώς θα μπορέσει να πλουστεύσει τους ελέγχους. Όχι μόνο για τις ε, κρατικές και ενισχύσεις, αλλά και για κάποιες ε, προσαρμογές που δεν ζητούνται για τις άμεσα κονδύλια, για τις άμεσες πληρωμές. Θέλω να συμφωνήσω με τον κύριο Πόμπης για το ε, πόσο σημαντικά είναι κάποια πράγματα που ανέφερε. Νομίζω ότι η αιρεσιμότητα εξάντε είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πραγματικά αυτό μας βοηθά στην έγκαιρη διάγνωση. Και θέλω να πάρω σε ένα παράδειγμα πολυπλοκότητες ε, και το πλαίσιο του performance fair και εμείς ε, έχουμε δημιουργήσει ε, ουσιαστικά ένα μηχανισμό για να αξιολογήσουμε το στρατηγικό πλαίσιο. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό γιατί ήταν πολύ σοφός ο κανονισμός, θέσπισε κανόνες, πρόβλεψε κανόνες και για να αξιολογήσουμε αυτό το μέσο κατά τη διάρκεια της όλης άσκησης. Έτσι λοιπόν πρέπει να έχει πραγματική εφαρμογή που να μας οδηγεί όλο και πιο κοντά στα αποτελέσματα και να μην και επικεντρωνόμαστε μόνο στη συμμόρφωση και να μην κάνουμε το σύστημα μόνο ένα σύστημα δεσμευτικό ο κανόνας νη 2, συν 3 εγγυάται ότι δεν μπορεί κάποιος να βάλει κατά μέρου κονδύλια χωρίς να τα δαπανίσει, γιατί αν δεν δαπανηθούν επιστρέφονται το ποσό που δεν ανήκει στη χρηματοδότηση Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτού. Σε ό,τι αφορά στα λάθη, που προκύπτουν από αυτό το όλο το κοραστικό εγχείρημα, τα κράτη-μέλη πρέπει να καλύψουν πόρους ε, που είχαν δαπανίσει και που ουσιαστικά ε, δεν θα αποζημιωθούν για αυτές. Yeah, vielen Dank. Das Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η εισαγωγή αυτή για την ε, στήριξη που ζητεί και τις διορθώσεις ε, που πρέπει να γίνουν. Ε, χαιρόμαστε πολύ και περιμένουμε να δούμε και τη συνέχεια. Τώρα τη συνέχεια η κυρία Τόαντερ, Γενική Γραμματέα στο Υπουργείο για τα Κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Ρουμανία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Καλώς ήρθατε κιόλας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε σήμερα εδώ. Ίσως η κατάσταση να μην είναι η πιο απλή γιατί έχει κατονομαστεί η Ρουμανία εδώ και δεν είναι εύκολο να έχετε κανείς εδώ και να πρέπει να αναγνωρίζει τα ασφάλματά του. Πάντως είναι καλή αυτή η ανταλλαγή απόψεων ε, και μάλιστα με αυτούς που είναι οι πιο καλοί μαθητές. Και έχουμε ανταλλαγή απόψεων για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε εμείς οι ουραγοί, οι τελευταίοι. Με εξαίρεση βέβαια ότι είναι Κροατία. Είναι καλό επίσης να διδαχθούμε ένας από τον άλλο πάνω στο τι πήγε καλά και ιδίως πάνω στο τι δεν πήγε καλά. Οπότε έτσι θα μπορούσαμε ίσως να προσαρμοστούμε και να απλουστεύσουμε τα πράγματα. Γιατί η Ρουμανία περίοδος 2007-2013 <clears throat> ήταν η πρώτη ε, διαδικασία στην οποία συμμετείχαμε. Είχαμε μόνο την προενταξιακή εμπειρία, τα κονδύλια τα προενταξιακά. Όχι ότι αυτό δεν ήταν χρήσιμο, αλλά δεν μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε, επειδή ήταν τελείως διαφορετικοί οι κανόνες που ίσχυαν προένταξης και μετά την ένταξη. Για πρώτη φορά λοιπόν είχαμε να αντιμετωπίσουμε τους κανόνες της πολιτικής συνοχής. Η Ρουμανία επίσης έχει και ένα ειδικό καθεστώς αν θέλετε, γιατί είμαστε επιλέξιμοι και για το Ταμείο Συνοχής που χρηματοδοτεί ευρείας κλίμακας υποδομές, ε, project ε, μεγάλης κλίμακας ε, και με μεγάλο χρονικό ορίζοντα και δεκαετία ακόμη. Και αυτό καθιστά πολύ δύσκολο το να μπούμε στο νη 1, νη 2, νη 3 ή και από την αρχή ακόμα. Όπως είπα λοιπόν και στην αρχή, η Ρουμανία είναι δύσκολη. Το ποσοστό απορρόφησης βέβαια έφτασε το 90% που μπορεί και να μην είναι η καλύτερη θέση, μπορεί να έχουμε φτάσει, αλλά είναι ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα. Γιατί αρχικά ήμασταν στα επίπεδα του 7% το 2009. Άρα έχουμε επιταχύνει, κάναμε ό,τι το δυνατόν και νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό έχουμε καταφέρει να πιάσουμε ρυθμό και να επιταχύνουμε στην υλοποίηση και να βοηθήσουμε και τους δικαιούχους μας, διότι ναι, πράγματι το θέμα είναι ο έλεγχος, είναι η απορρόφηση, οι κανόνες, όμως οι πιο σημαντικοί παράγοντες και πρωταγωνιστές της πολιτικής συνοχής είναι οι δικαιούχοι και αυτοί ακριβώς θα πρέπει να λάβουν την απαιτούμενη υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υλοποίησης. Βέβαια το τελικό ποσοστό απορρόφησης ε, θα είναι γνωστό όταν έχει γίνει ο έλεγχος ε, και η εξέταση της τελικής δήλωσης. Ωστόσο, ελπίζουμε το 90% που έχουμε ήδη δηλώσει στην Κομισιόν να σταθεροποιηθεί και να είναι λίγο πολύ το τελικό ποσοστό απορρόφησης. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πέραν των δαπανών που δηλώσαμε στην Κομισιόν, αντιμετωπίσαμε ένα ακόμη πρόβλημα, που ήταν δημοσιονομική διόρθωση, που στο τέλος για τη Ρουμανία έφτασε τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Και βγήκαν από το κρατικό προπολογισμό αυτά τα χρήματα ή από του τελικού δικαιούς αναλόγω του είδου των δικαιούχων για του οποίου συζητούσα Α, κατά περίπτωση. Αυτό το αποτέλεσμα όπως μπορεί και να μείνει το καλύτερο δυνατόν. Για εμάς όμως, που ήταν η πρώτη δημοσιονομική τέτοια άσκηση, μας δίνει τη δυνατότητα τώρα να μελετήσουμε και αυτά που κάναμε λάθος και αυτά που κάναμε σωστά και να αντλήσουμε τα διδάγματά μας επί δημοσιονομικής κρίσης νομίζω ότι καταφέραμε να κάνουμε πάντως κάποια πράγματα και τι διδαχθήκαμε μεταξύ άλλων. Πρώτον, ιδίως ό,τι αφορά τα project μεγάλης κλίμακας που είμαστε δικαιούχοι όπως είπα και από τα κοντιλεκτομείου συνοχής. Μια από τις σημαντικές ανάγκες της Ρουμανίας που παραμένει είναι οι υποδομές. Μπορεί να ήμασταν οι πρώτοι που ε, είχαμε την περιοδο 2017 2007-2013 τα πρώτα εγκεκριμένα project και από τις πρώτες χώρες για τις οποίες εγκρίθηκαν και τα προγράμματα και το σύστημα διαχείρισης, πάντα για την περιοδο 2017-2013 το στρατηγικό πλαίσιο, εγκρίθηκε το νέο του 2007. Παρ' όλα αυτά, σε ό,τι αφορά την υλοποίηση, είμαστε τελευταίοι. Και αυτό δεν σημαίνει ότι ο δικαιούχοι μας δεν ξέρουν τι χρειάζονται. Ούτε σημαίνει ότι εμείς δεν ξέρουμε στη Ρουμανία τι θέλουμε και τι χρειαζόμαστε ή δεν κάναμε ε, την εργασία που έπρεπε να γίνει για την ανάλυση των αναγκών. Το θέμα είναι ότι σε μεγάλα project, μεγάλες κλίμακες project, πολλές φορές χρειάζεται πολύ καλή προετοιμασία και μακροχρόνια προετοιμασία. Σε αυτή την κούρσα ε, και για την αύξηση της απόρροφησης και για να μην χάσουμε χρήματα στον, με το κουμπά στο κανόνα συν 2 συν 3. Κάποιες φορές, κάποια συγκεκριμένα project δεν, τα δεν προετοιμάστηκαν σωστά, δεν δόθη ο πετούμενο χρόνος για να μελετηθεί η ποιότητα και η ποιότητα των μελετών σκοπιμότητας δεν ήταν ίσω η καλύτερη δυνατή, γιατί πάντα λέμε ότι πρέπει να ανατεθούν τα κονδύλια εκεί και να υπογραφούν οι συμβάσει και τα λοιπά, γιατί θα τα χάσουμε τα χρήματα. Άρα βιαζόμασταν λίγο σε κάποιε περιπτώσει και αυτό ήταν ένα από τα βασικότερα προβλήματα. Δηλαδή, τα μεγάλα σχέδια στον τομέα των υποδομών δεν ήταν σωστά προετοιμασμένα και σε συνεργασία με τους δικαιούχους. Επίσης, δεν είχαμε την ε, δρεωμένη διοικητική ε, ικανότητα που θα μας επέτρεπε να διαχειριστούμε τα μεγάλες κλίμακες αυτά ε, σχέδια. Γιατί πρέπει να το παραδεχτούμε, άλλωστε είναι και πολύπλοκοι οι κανόνες, οι ευρωπαϊκοί, και έρχονται να προσθεθούν και στους ήδη πολύπλοκους εθνικούς κανόνες που δυσκολεύουν ακόμη πιο πολύ τα πράγματα για τους δικαιούχους μας. Αυτή ήταν μια από τις αιτίες λοιπόν που οδήγησε στα χαμηλά ποσοστά φυσικά στον τομέα των μεταφορών, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα μεταφορών ξεκινήσαμε να χρησιμοποιούμε την τεχνική συνδρομή που παρέχει ιδίω η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυξήσαμε επίση τι επαφέ με το Jaspers και τη συνεργασία μας. Θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες της Κομισιόν γιατί μπορεί να μην σε με τον σωστό τρόπο, αλλά ε, μας συμπεριέλαβε σε αυτό το διάλογο. Και κάτι από τα καλύτερα ίσως ήταν η εξάντε αιρεσιμότητα ε, της μεταφορές. Γιατί έτσι και εμείς και οι δικαιούχοι αρχίσαμε να σχεδιάζουμε, να προγραμματίζουμε μασοπρόθεσμα και, και μακροπρόθεσμα. Ένα άλλο θέμα για το οποίο παρατηρούνται, λόγω το οποίο παρατηρούνται αυτά τα προβλήματα είναι η χρηματοπιστωτική κρίση. Το πρόβλημα της ταμιακής ροής ε, και του κρατικού προπολογισμού. Το είπε και η Ταλίδα συνάδελφος Πρώτα απ' όλα, δικό μα καθήκον σε εθνικό επίπεδο είναι να πληρώσουμε του δικαιούχου μα. Αν δεν του πληρώσουμε, δεν μπορούμε να ζητήσουμε χρήματα από την Επιτροπή. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε επιστροφή χρημάτων. Το 2008-2009, που η Ρωμανία χτυπήθηκε σκληρά από τη χρηματοπιστωτική κρίση, είχαμε πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμή των δικαιούχων. και μεγάλος τζίρος προέκλειθη για τη διοίκηση. Υπήρξαν όμως περικοπές και κάποιοι έφυγαν από τη διοίκηση. Και υπήρχε το πρόβλημα το επίπεδο της ταμιακής ροής. Δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν τους ίδιους πόρους στα σχέδια. Πήραμε τα μέτρα μας χρησιμοποιούμε ακόμη το χρηματοοικονομικό αυτό μηχανισμό. Στηρίξαμε τους δικούς ουσιαστικά για την πληρωμή των τιμολογίων από τον κρατικό προϋπολογισμό για να μην συνεισφέρουν το συνολικό ποσό από το δικό τους προϋπολογισμό. Μας καταθέτουν δηλαδή το τιμολόγιο, ελέγχουμε και τους δίνουμε έπειτα τα χρήματα. Και παίρνουμε αυτό το ρίσκο, αν μπορώ να το πω έτσι, και αυτό ίσω είναι και ένα πρόβλημα, παίρνουμε ένα ρίσκο πάνω στον κρατικό προπολογισμό, πληρώνοντα από τον κρατικό προπολογισμό. Αυτό ο μηχανισμό ήταν δύσκολο να τεθεί σε λειτουργία, ιδίω με το Υπουργείο Δημοσίων Οικονομικών και παρά τι διασφαλίσει που ζητούνται πάντοτε από τα Υπουργεία Δημοσίων Οικονομικών ε, για τους δημόσιους πόρους πάντα. Πάντως το σύστημα αυτό τώρα έχει τεθεί σε λειτουργία και μειώθηκε ε, ο χρόνος από την αξίωση, το αίτημα της πληρωμής μέχρι την πληρωμή σε 20 μέρες. Μέσα σε 20 μέρες, λέει το πολύ, ε, πληρώνονται οι δικαιούχοι όταν υποβάλλουν το αίτημά τους. Ένα άλλο πρόβλημα που είχαμε και ελπίζουμε να έχει λυθεί πια, είναι ο συντονισμός δεν υπήρχε συντονισμός σε κεντρικό επίπεδο σε σχέση με τις αρχές που δεν χειρίζονταν τα κονδύλια της Ένωσης. Δεν υπήρχε κεντρικός φορέας συντονιστικός που να καθοδηγεί και να δημιουργεί αυτό το πλαίσιο, αυτό το περιβάλλον ασφαλείας, αν μπορώ να το πω έτσι, που συνέδεε τους ε, ενδιάμεσους και τους δικαιούχους. Γι' αυτό λοιπόν το Υπουργείο ε, Νοσιακών Κονδυλίων από κοινού με το Υπουργείο Περιφερικής Ανάπτυξης ε, συνεργάζονται, έχουν την ίδια λογική ε, παρέμβαση, αν θέλετε, οι διαχειριστικές αρχές στο σύνολό τους πλέον πάγονται στο δικό μας Υπουργείο. Άρα μπορούμε να έχουμε οριζόντιους κανόνες, οριζόντια προσέγγιση και οριζόντια εφαρμογή διότι υπήρχαν διαφορές στην υλοποίηση. μεταξύ ας πούμε του περιφερειακού περιφερειακού προγράμματος και της ανταγωνιστικότητας. Και το τελευταίο και πιο σημαντικό είναι η υποστήριξη που παρέχουμε στους δικαιούχους μας. Δεν συμφωνώ ότι δεν ξέρω τι να κάνουμε τα χρήματα. Δυστυχώς επειδή συζητήθηκαν λιγότερο επίγονες περιοχές, εμείς έχουμε 7 στις 8 περιφέρειες σε αυτή την κατηγορία. Πολύ χαμηλή διοικητική δυνατότητα. Πρέπει να αποστηριχθούν. Πολλές είναι οι ανάγκες. Αλλά χρειάζεται στήριξη από τις αρχές, όχι τις εθνικές μόνο, αλλά και τις ευρωπαϊκές. Είναι απαραίτητη αυτή η υποστήριξη για να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε όλους τους πόρους που είναι απαραίτητη και να πετύχουμε τους στόχους της πολιτικής συνοχής για να μην είμαστε πίσω. Γι' αυτό και θεωρώ ότι αυτή η πρωτοβουλία για τις ε, περιοχές που έχουμε μείνει πίσω, τις μενεκτικές περιοχές, lagging regions, πρέπει να υποστηριχθεί. Υπάρχουν πολύ απλές πλέον προτάσεις, άρα κινούμαστε πολύ γρήγορα. Τις συζητούμε τις προτάσεις αυτές με όλους τους εμπλεκομένους φορείς και στη Ρουμανία τώρα παρέχουμε τα κονδύλια για να ξεκινήσει η χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ. Η πρωτοβουλία της ευφυού εξειδίκευσης, αν μπορώ να την πω έτσι, σε επίπεδο περιφερειών. Και με βάση τα αποτελέσματα που θα έχει αυτή η πρωτοβουλία, ελπίζω να αρχίσουμε και με τις άλλες έξι. που δεν είναι τόσο ανεπτυγμένες το Βουκουρέστι μόνο λοιπόν, αναπτυγμένη που είναι σαν ε, το φωτεινό αστέρι που φωτίζει όλους τους άλλους. Μπορεί να μην είμαστε πρωταθλητές στην απορρόφηση, τα αποτελέσματα όμως που πέτυχε η Ρουμανία χρησιμοποιώντας ε, την πολιτική συνοχή, νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να αναγνωριστεί. Έχουμε φτιάξει δρόμους, έχουμε εκπαιδεύσει κόσμο, έχουμε μειώσει την ανεργία, έχουμε στηρίξει τις ΜΜΕ ιδίως σε πάρα πολύ δεινούς καιρούς, όπως ήταν ε, ο καιρός της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά πρέπει να εκτιμήσουμε την ε, σπάρεμπά σας ε, Γιατί πρέπει να ξεπέντε σωστά τα κόντυλα, γι' αυτό είστε κι εσείς άλλωστε εκεί. Να δώσω τώρα το λόγο για ερωτήσεις στον κύριο Πυρίνσκι. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι και τρεις παρουσιάσεις πάνω κάτω επιβεβαίωσαν αυτό που προσπάθησα να τονίσω αρχικά. Υπάρχουν παραδείγματα χωρών που είναι ιδιαίτερα επιτυχής στην απορρόφηση κονδυλίων. Ανέφερα τα ποσοστά των πληρωμών που έγιναν το 2016 ως ποσοστό των αρχικών προβλέψεων που έκανε οι χώρες και στην περίπτωση χωρών όπως η και Φιλανδία αυτές οι απαιτήσει ήταν υψηλότερε από τα αρχικά προβλεπόμενα στη Σουηδία κατά 93%. Άλλες χώρες ήταν σχεδόν ανίκανες να καταθέσουν μια τέτοια απέτηση για πληρωμή 6% για την Κροατία. Η Ρουμανία φαίνεται έχει πολλή δουλειά ακόμα για να καταθέσει να εισαγάγει μια τέτοια απέτηση πληρωμών ως ποσοστό των πληρωμών που είχαν προβλεφθεί. Βέβαια και η δική μου χώρα αντιμετωπίζει μια σειρά προβλημάτων που έχουν να κάνουν με την ε, επιτυχία απορρόφηση. Τώρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε όλο αυτό το εγχείρημα, δηλαδή η απορρόφηση, έχει να κάνει με το στόχο της ε, μεγαλύτερης συνοχής και της πρόθεσης της σύγκλησης. Δηλαδή, το να κάνουμε διάφορε μελέτε και να δείχνουμε ότι κάποιοι είναι επιτυχεί, ενώ άλλοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, δεν απαντά το ερώτημα ποια είναι τα κατεπήγοντα μέτρα που μπορούν να ληφθούν από την Κομισιόν για να ευθυγραμμιστούν περισσότερα αυτά τα ποσοστά. Και πιστεύω ότι όπως αναφέρθηκε αυτό είναι ένα πρόβλημα στο σύστημα. αναφέρθηκε από κάποιους ομιλητές αναφέρθηκαν και στα πορίσματα του ελεκτικού συνεδρίου στην καθυστερημένη έγκριση και των κανονισμών αλλά και του δημοσιονομικού πλαισίου που οδήγησε στην εξή κατάσταση. Στα δύο πρώτα έτη της περίοδου αυτής, 2015 και 2016, να είναι χαμένα χρόνια για την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Επίσης πιστεύω ότι όσο ακούσαμε από την Κομισιόν στη δεύτερη παρέμβαση, μας οδηγεί σε ένα πιθανό συμπέρασμα ότι έχουμε εντοπίσει μια σειρά συμφορήσεων σε ό,τι αφορά την πιο επιτυχή και εύκολη απορρόφηση. Γιατί από ό,τι ακούσαμε έχουν ε, υπάρξει καθυστερήσεις ε, στη βελτίωση των ε, σχεδίων. Και ακούσαμε και τον εκπρόσωπο της Γαλλίας, ο οποίος μας τόνισε την ανάγκη να είναι κανείς γρήγορος, ταχύς. Και πολλές φορές το βέλτιστο είναι χειρότερο του καλού, είναι ο εχθρός του καλού. Έτσι λοιπόν πρέπει να βρούμε μια πολύ προσεκτική ισορροπία μεταξύ του έλεγχου, του επαναλέγχου, πριν την έγκριση και να προχωρεί κανείς. Και φυσικά θα πρέπει κανείς να παρακολουθεί την όλη διαδικασία και να διασφαλίσει, να είναι σίγουρος ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι για παρατυπίες, για πάτες κτλ. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου οι καθυστερήσεις επαναλαμβάνονται. Αναμέναμε μια πρόταση της Κομισιόν για ένα πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο μέχρι το τέλη αυτού του έτους και καταλαβαίνουμε ότι ίσως κάτι τέτοιο μάλλον θα γίνει περί τα μέσα του επόμενου έτους. Η Κομισιόν ανέφερε το 7ο φόρουμ για τη συνοχή που έλαβε χώρα όμως δεν μας έχει δώσει την 7η έκθεση για τη συνοχή κομισιών. Κάτι που έπρεπε να γίνει πριν τρία χρόνια, όταν είχε προετοιμαστεί πολύ καλά αυτό το φέρου μέσω μιας ε, πλήρους έκθεσης που ακριβώ μας έδειχνε το επίπεδο της συνοχής που είχε επιτευχθεί και τις προκλήσεις. Πολύ ωραίες δύο ημέρες συζήτηση, ωραίες οι ομιλίες που ακούσαμε, αλλά δεν μπορούσαμε να εξετάσουμε εις βάθος ποιες είναι οι προκλήσεις για να προχωρήσουμε με τη συνοχή. Επίσης, θα ήθελα να καλωσορίσω τις τρεις παρουσιάσεις ε, και να πω ότι νιώσα μια ικανοποίηση με τις παρουσιάσεις που ακούσαμε, όμως από την άλλη πιστεύω ότι η Κομισιόν μπορεί να πετύχει μια ακόμη καλύτερη διαδικασία απορρόφησης. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Έχω και εγώ ερωτήσεις. Η κυρία από την Ιταλία. Θα είπα πολύ ξεκάθαρα και εύκολα σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση. Μας δείξατε κάποια ε, διαγράμματα για τη ρύθμιση. Φαντάζομαι θα πρέπει να τοποθετηθεί και η Κομισιόν. Γιατί πηγαίνει, βλέπω, πολύ προς τα πάνω ε, το διάγραμμα σε σχέση με τη ρύθμιση και αυτούς τους κανόνες. Θα ήθελα να μας πείτε κάποια πράγματα. Γιατί μιλάμε συνέχεια για την απλούστευση. Ας καταλάβουμε πρώτα τι θα πει απλούστευση, δηλαδή κατευθυντήριες γραμμές, αν μπορείτε να μας το απαντήσετε αυτό και για την εκπρόσωπο πάντα από την Ιταλία. Έχουμε την ε, Καμπανία, την Σικελία και την Τρίτη και την Κατάμπρια. Για το 2010-2011 εκεί πήγαμε στην Καμπανία, πριν δύο χρόνια πήγαμε στη Σικελία. Και πραγματικά, επειδή η Ιταλία είναι κεντρωτικό μέλος ε, της Ένωσης, ε, μας ε, φάνηκε το ότι υπάρχουν αυτά τα σοβαρά περιφερειακά προβλήματα. Πήγαμε εκεί, μιλήσαμε με πολλούς και δεν είχαμε πολύ καλή εντύπωση. Γιατί δεν φαίνεται να γίνονται πολλά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Τι νέα έχετε για τη βελτίωση της απορρόφησης μέσω των μέτρων τα οποία έχουν πάρθει και για την πρόσωπο της Ρουμανίας. Αναγνωρίσατε τη δυσκολία. Είναι μια χώρα που ακόμα έχει πάρα πολλά προβλήματα μετά από 10 χρόνια. Είπατε ότι έχει μειωθεί η διοίκηση, όγκος της διοίκησης. Έχουν φύγει πάλι. Πολλέ φορέ όταν αλλάζει κυβέρνηση, αλλάζει τελείω, ανακυκλώνεται τελείω και το ε, διοικητικό προσωπικό. το ίδιο συμβαίνει και στη Ρουμανία. Αλλάζεται τελείω ε, δηλαδή και το προσωπικό στα Υπουργεία. Και τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στην ε, Ρουμανία. Για τον Δανό, δυστυχώς δεν έχω κανένα ερώτημα, λυπάμαι γιατί είναι τόσο καλά τα πράγματα, μας εντυπωσιάσατε. Ίσως ένα θέμα είναι ο διοικητικός φόρτος, αυτά τα έγγραφα. Εσείς πώς θα καταφέρετε καλύτερα σχέση με άλλους για τους οποίους είναι μεγάλο πρόβλημα όλο αυτό το χαρτομάνι. Ο κύριος Πόπενς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να φύγω σε 10 λεπτά. Ελπίζω να μην σας ε, πειράζει αυτό. Είχα προγραμματίσει να μείνω εδώ μέχρι τις 5. Οι συνεργάτες μου θα μείνουν. Ήθελα όμως να επιβεβαιώσω ότι συνεργαζόμαστε πολύ στενά με όλα τα κράτη-μέλη. Πράγματι. Και επίσης το επίπεδο διοικητικής δυνατότητας διαφέρει είπατε κι εσείς για τις περιφέρειες και εμείς δημοσιεύουμε μια έκθεση και ξέρουμε ότι η στενοπός. Δεν εξαρτάται από μένα για να αντιμετωπιστεί. Είναι θέμα διακυβέρνησης, έχει σχέση με ε, θέματα παιδείας, ε, αγοράς εργασίας, που δεν είναι αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε και τα οποία κάνουμε ιδίως για να βοηθήσουμε συγκεκριμένες περιφέρειες. Πράγματι, ε, όσον αφορά τις ε, αρχές της Δανίας, έγιναν σοβαρές διαπραγματεύσεις αλλά πολύ αποτελεσματικές. Και αυτό πριν καν ξεκινήσει η περίοδος. Είναι, γίνεται. Αυτό που σημαίνουν όλα αυτά είναι ότι πράγματι οι καταστάσεις διαφέρουν, μερικές είναι δύσκολες, προσπαθούμε να συνεργαστούμε με κάθε περιφέρεια όπως είναι δυνατόν. Η, η Κομισιόν δεν αποτελεί τη στενοπό στην υλοποίηση μπορούμε να το συζητήσουμε. Η καθοδήγηση σκοπό έχει την παροχή ασφάλειας δικαίου. Μην φανταστείτε ότι είναι θέμα μόνο καθοδήγησης. Μα ζητούν την καθοδήγηση στα κράτη-μέλη. Μπορώ να εξηγήσω γιατί το κάνουν και ταυτόχρονα επικρίνουν το, την υπερβολική καθοδήγηση. Αυτό το πατήσουν οι Μα το θέμα δεν είναι η ορολογία. Υπάρχει κάτι που προσπαθούμε να κάνουμε με όλους. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται στην τρέχουσα περίοδο, όπως η απλούστευση του κόστους. Είναι πράγματα που γίνονται εύκολα, αλλά που δεν τα εντοπίζουν. Οι αρχές. Δεν είναι μόνο θέμα ορολογίας, είναι και θέμα ε, του τι έχει γίνει πίσω από εκεί. Αποτελέσματα. Δεν είναι μόνο η προσήλωση στα αποτελέσματα, είναι ένα ολόκληρο πλαίσιο επιδόσεων που έχουμε δημιουργήσει και πρέπει να το σεβόμαστε. Το επίπεδο προγραμματισμού είναι πολύ διαφορετικό. Υπάρχουν εθνικά προγράμματα με πολλά, για όλα τα ταμεία που καλύπτουν όλη τη χώρα και υπάρχουν περιφερειακά συγκεκριμένα προγράμματα που, που ε, καλύπτουν μια συγκεκριμένη περιοχή. Όλοι χρειάζονται αποτελέσματα και δείκτες. Όλα αυτά θα συνεχίσουμε να τα κάνουμε. Όταν μιλάω για το μέλλον αυτής της πολιτικής και πάλι ε, θα αναφερθώ στον εκπρόσωπο της Δανίας. Αυτή ήταν η προσέγγιση μας εκεί. Δεν αναφερθήκαμε σε φακέλους, είπαμε ανάγκες, πώς μπορούμε να, τους, να τις καλύψουμε και μετά από ένα μήνα θέσαμε προτεραιότητες και προσπαθήσαμε να τις επιδιώξουμε. Και αυτό κάνουμε και σε αυτή την περίοδο. Η ευελιξία δεν σημαίνει ότι ο καθένας δουλεύει ό,τι ώρα θέλει, αλλά ε, η χρηματοδότηση ε, προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η, η τρομοκρατία έχει επηρεάσει τους πολίτες αυτό, δεν ήταν κάτι που είχε ληφθεί υπόψη διαπραγματεύσει, αλλά τώρα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν μιλάμε για χρηματοδότηση και έχουμε δώσει μια προτεραιότητα για στη μετανάστευση, γιατί μακροπρόθεσμα πιστεύουμε ότι μέσω της ενσωμάτωσης μπορούμε να βοηθήσουμε και σε αυτό το τομέα. Έτσι λειτουργούμε και έτσι θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με συνεργασία με όλους τους εταίρους μας, ολόκληρη την Ευρώπη, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με το Ελεγκτικό Συνέδριο και πολύ σωστά. Επισημάνατε ότι το να υπάρχει έλεγχος επιδόσεων στα αεροδρόμια κάνουμε το βασικό τεν δέκα. Και δεν ασχολούμαστε με τα μικρά πράγματα που ενδεχομένως χρειάζονται. Ε, κάνουμε πολλά για την εκ των προτέρων ρεσιμότητα. Ε, και ευχαριστούμε τη Ρουμανία που είπε ότι αυτό ήταν απαραίτητο. Το ίδιο χρειάζεται και σε άλλους τομείς. Συνεργαζόμαστε με τα κρατημέλη για να τα συμπεριλάβουμε. Και εγώ ζητώ να αναγνωριστεί το έργο της Επιτροπής στην όλη αυτή διαδικασία γιατί πιστεύω ότι έχουμε φτάσει στο διάστημα που μπορούμε πλέον να, να χτίσουμε για μετά το 2020. Αυτό πρέπει να τεκμηριωθεί με στοιχεία, το προσπαθούμε στο τέλος χρονιάς. Θα υπάρχει μια στρατηγική έκθεση που θα στηρίζεται από τις, στις εκθέσεις των κρατών μελών, τις διαχειριστικές αρχές. Η έκθεση συνοχής ε, καθυστέρησε σκοπίμως γιατί πάντοτε μας κατηγορούσαν ότι τις, θέλουμε εκ των προτέρων και μετά γίνεται εκ των υστέρων συζήτηση. Τώρα περιμένουμε το αντίστροφο, να ακούσουμε τι έχουμε να, ε, να λάβουμε, αυτά που έχουμε να λάβουμε και μετά να συντάξουμε. Και μετά ε, θα έχουμε την έκθεση πρόοδου κομισιών για όλα τα διαρθρωτικά ταμεία. Θα δούμε και τα διάφορα στοιχεία. Θα έχουμε έκθεση για τις ε, περιοχές που καθυστερούν, ε, για την εξυπνή εξειδίκευση. Θα έχουμε μια άλλη έκθεση αργότερα φέτος και σκεφτόμαστε το μέλλον με πολύ δραστήρια. Αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο επί του μέλλοντος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Ähm, Ευχαριστώ. Καλές, ε, καλό κουράγιο και καλή διασκέδαση και στη συνέσεια για την ε, γάμα δέλτα Εσείς παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, δύο ερωτήσεις μου έγιναν νομίζω. Πρώτον, αλλά θα ήθελα να κάνω μια σύντομη παρατήρηση για το θέμα του προσωπικού που αναφέρατε εσείς κυρία Πρόεδρε. Μπορώ να επιβεβαιώσω και όλοι όσοι συνεργάζονται με τα διαρθρωτικά ταμεία και τον κανονισμού, τους κανονισμούς όλα αυτά τα χρόνια θα το επιβεβαιώσουν αυτό. Κάτι που είναι σημαντικό είναι ότι το προσωπικό πρέπει να είναι έμπειρο και να ασχολείται, να έχει προσήλωση προς την υλοποίηση. Αυτό το έγραψα και στις διαφάνειες και αυτό έχει δείξει και η εμπειρία μου και από πλευράς και από πλευράς Επιτροπής και από πλευράς Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με τα χρόνια, ακόμα και την εποχή που ήμασταν πολύ μικροί, είχαμε αυτή την εμπειρία και έμπειρο προσωπικό που είχε σκοπό την υλοποίηση. Δεν ζηλεύω την κατάσταση κρατών μελών όπου για διάφορους λόγους πρέπει να αλλάζουν το προσωπικό τους από το ένα διάστημα στο άλλο. Εμείς διατηρούμε τους ίδιους. Τώρα, για ποιο λόγο ο κανονισμός γίνεται όλο και ογκοδέστερος. Εν μέρη θα συμφωνήσω με τον κύριο Πόπενς. Εμείς μερικές φορές τα κράτη-μέλη ζητάμε περισσότερες οδηγίες συγκριτικά ή σε επίπεδο επιτροπής. Ζητάμε προβλεψιμότητα ή ε, εξηγήσεις για έναν κανονισμό που δύσκολα είναι κατανοητός ή καμιά φορά εμείς ε, έχουμε ένα αποτέλεσμα σε σχέση με μια κατευθυντήρια γραμμή. Αυτό δεν θεωρώ ότι είναι πολύ ορθολογικό από πλευράς κρατών μελών. Μερικές φορές και εμείς πρέπει να πάρουμε τον κανονισμό ως έχει χωρίς κατευθυντήριες γραμμές, χωρίς λεπτομερείς επεξηγήσεις επιπλέον των όσων λέει ο κανονισμός. Το λέω αυτό ως μικρό κράτος μέλος. Υπάρχει μέρος του κανονισμού που δεν το χρησιμοποιώ. Δεν χρησιμοποιώ τον κανονισμό που αφορά τα μεγάλα έργα υποδομής, γιατί δεν τα κάνουμε εμείς αυτά. Άρα δεν έχω τέτοιο θέμα. Υπάρχει ένα κομμάτι του κανονισμού που το ε, παρε, αντιπαρερχόμαστε. Αλλά δουλεύουμε με τον κανονισμό και του επιτιθέμεθα. Δηλαδή, το θεωρούμε κομμάτι της ζωής. Αυτό έχουμε, αυτό μας δώσανε και με αυτό θα δουλέψουμε αν πρόκειται η δαπάνη να γίνει σωστά, θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες. Αυτό το έχουμε δεχτεί, αυτό το έχουμε υποσχεθεί. Υπάρχει μέσα στα θεσμικά όργανα μια ε, κοινή διαχείριση και αυτό πρέπει να κάνουμε. Απλώς θα ασχοληθούμε περισσότερο με το να τον εφαρμόσουμε παρά με να τον συζητάμε τον κανονισμό. Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο μπορώ να περιγράψω την καθημερινή δουλειά μας. Μια σύντομη, σύντομο σχόλιο θα ήταν ότι η διαφορά ανάμεσα σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα χρηματοδότηση και το ένα εθνικό σύστημα, τουλάχιστον δικό μας, είναι ότι υπάρχουν διάφορα επίπεδα ελέγχου στο ευρωπαϊκό σύστημα ενώ στο εθνικό ε, σύστημα κυρίως έχουμε να κάνουμε με το Εθνικό Ελεγκτικό Συνέδριο. Και αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, εμείς, εμείς με τρόπο προβλέψιμο και σύμφωνα με τους κανόνες πρέπει να ανταποκριθούμε στις ανάγκες κάποιων ελέγχων. Η κατάσταση όμως έχει βελτιωθεί σύν το χρόνο γιατί ο έλεγχος έχει γίνει περισσότερο μια διαδικασία μάθησης και συγκέντρωσης. Σήμερα ο διάλογος που έχουμε με όλους τους ελέγχους και με την Επιτροπή για μας εμάς μας έχει επιτρέψει να χειριζόμαστε σωστά τον κανονισμό. Παραδείγματος χάρη, ο κανονισμός αναφέρει στον καθορισμό των αρχών. Στην περίπτωσή μας, ο καθορισμός των αρχών ήταν μια δικασία που ξεκίνησε για να εγκριθεί και να διοριστεί μια διαχειριστική αρχή η οποία διαχειρίζεται τα ευρωπαϊκά κονδύλια από το 1990. Αισθανόμαστε μερικές φορές ότι ο κανονισμός δεν εξυπηρετεί τους πάντες, αλλά τον σεβόμαστε ως έναν ευρωπαϊκό κανόνα, όπως οφείλουμε. 20 Είστε όμως ε, όλα αυτά τα 20 χρόνια πάντα στην κορυφή και ταυτόχρονα έχετε συλλέξει τελάχιστα εμπειρία. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στις επόμενες δύο μιλήτρες. Πρώτα η κυρία Τοάντερ και μετά η κυρία Γκρό. Ευχαριστώ πολύ σε ό,τι αφορά τον... Σε ό,τι αφορά τους ε, ορισμούς, ε, εγώ ε, ήδη ασχολούμαι με τη δημοσιοδίκηση. Ασχολούμαι με τη δημοσιοδίκηση εδώ και 15-16 χρόνια. Τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε σχετίζονται κυρίως από το 2009. Οι μισθείς, ε, όλη τη δίκηση, ε, έγιναν κάποιες περικοπές, γύρω στο 20%. Έτσι λοιπόν οι καλύτεροι, για να το πούμε έτσι, έφυγαν και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τους επαναφέρουμε. Δεν υπάρχει αρκετή σταθερότητα, το γνωρίζουμε αυτό πολλές φορές και γι' αυτό ως τμήμα της ε, δράσης ε, της ερεσιμότητας ε, υιοθετήσαμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Αυτό το έχουμε ξαναθετήσει το 2015 και τώρα βρίσκεται στο στάδιο εφαρμογής μαζί με τον νέο κανονισμό για τις δεμίσιους επαλλήλους. Έτσι λοιπόν, να πούμε ότι η ερωσιμότητα εξάντια κατά κάποιο τρόπο μας βοήθησε για να δημιουργήσουμε ένα σύστημα για τους δημόσιους υπαλλήλους γενικά που δεν σχετίζεται μόνο φυσικά με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ευρωπαϊκά κονδύλια, έχουμε εισαγάγει ένα σύστημα αξιολόγησης ε, βάση του οποίου όλοι οι διαχειριστές ε, και όλοι οι υπάλληλοι αξιολογούνται δύο φορές το χρόνο με ένα σύστημα με δείκτες επιδόσεων. Αυτό το αναπτύξαμε με τη βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ε, όμως ε, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το αναπτύξαμε κυρίως εμείς στο Υπουργείο Ευρωπαϊκών Κονδυλίων. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε αν κάνουμε τη δουλειά μας. Βέβαια, οι δείκτες των επιδόσεων ε, δεν μπορούν να είναι πάντα ποσοτικοί, γιατί αν ε, παραδείγματο το σχάρι ε, θέλουμε να κρίνουμε έναν αρμόδιο για την έγκριση κονδυλίων και να δούμε πόσα χρήματα εγκρίνει, μπορεί να εγκρίνει τα πάντα για να πάρει τον πόνους του. Ενώ αν θέλουμε να ελέγξουμε πόσες παρατυπίες ε, μπορεί να εντοπίσει ένας ε, αρμόδιος στον τομέα αυτό, μπορεί να ε, βρίσκει παρατυπίες παντού για να λέει έκανα τη δουλειά μου. Τέλος πάντων έχουμε αυτό το πλαίσιο επιδόσιο και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που τώρα είναι η τρίτη χρονιά που το εφαρμόζουμε. Και φυσικά βλέπουμε αποτελέσματα σε επίπεδο διοίκησης. Βέβαια, εξακολουθούμε να έχουμε πολλά να κάνουμε για να εφαρμόσουμε την ε, διοικητική μεταρρύθμιση. Όπως σας είπα, έχουμε μια στρατηγική που θα πρέπει να εφαρμοστεί μέχρι το 2020 και πέρα από το 2020. Όμως ήδη έχουν γίνει συγκεκριμένα βήματα και θα έρθουν ε, και άλλα μέτρα προς εφαρμογή. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω, πρέπει να φύγετε καλή τύχη και καλή επιστροφή στη Ρουμανία. Οι συνάδελφοί μου θα παραμείνουν, λέει του το Άντα, και θα φύγουν το πρωί αύριο. Αν έχετε ερωτήσεις λοιπόν μπορούν να, να τις σημειώσουν και θα σας απαντήσουν το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρος. Ε, κυρία Αγκρό. Ευχαριστώ. Η ερώτησή σας ακριβώς έχει να κάνει με τους τρεις λόγους που ανέφερα για την περίοδο 2007-2013 δημιουργήσαμε μια ειδική task force στην Ιταλία και δημιουργήθηκε από την ίδια την περιφέρεια με τη στενή συνεργασία της Κομισιόν, η οποία πάντοτε μας βοήθησε. Βλέπουμε όμως ε, ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτές της Task Force. Ε, έκλεισε με απορρόφηση 104% ε, η Καλάβρια στο 109% είχε σημαντικό βερμπούκινηση και η Λία 96,7% δηλαδή είχε κάποια μικρή καθυστέρηση σε σχέση με το 100% όμως ε, είχε και ένα περιθώριο λάθος με 0,5% δηλαδή όλες οι διαδικασίες παρακολουθήθηκαν και είναι ε, πολύ πιο κάτω από το 2%. Τώρα, θέλουμε να δούμε τι γίνεται με το 2014-2020. Οι διαχειριστικές αρχές στην Καλαβρία και στη Σικελία μείναν οι ίδιες. Έχουμε δηλαδή σταθερότητα και έχουμε και τη γνώση, την τεχνογνωσία στην ε, Task Force. Και μπορέσαμε όλη αυτή την τεχνογνωσία να τη διατηρήσουμε εντός ε, των περιφερειακών δομών και τελικά όταν ε, μία μέθοδο την προσλαμβαίνει κάποιος αρχίζει τελικά να λειτουργεί για την ε, καμπανία μπορώ να σας πω ότι άλλαξε η διαχειριστική αρχή, αλλά όχι οι άνθρωποι που δούλευαν στην ίδια τη δομή και εκεί υπήρχε συνέχιση. Αν ε, δούμε τώρα την επιλογή των σχεδίων, που είναι ένας από τους δείκτες στην ε, έναρξη της προγραμματικής περίοδου. Και πρέπει να ξέρουμε ότι ο κανονισμός εγκρίθηκε το 2014 έτσι, λοιπόν, είχαμε και ένα χρόνο κενό σε σχέση με την έρεξη της περίοδου στη Σικελία. Ε, τα προγράμματα που επιλέχθηκαν για το 31% των φόρων στην Καλάβρια για το 35% και στην Καμπάνια για το 54%. Και αυτό γιατί ήρθε αυτή η τόσο σημαντική βελτίωση. Ίσως δεν δούμε ακόμα τις πληρωμές, αλλά υπάρχει ένας λόγος. Δεν υπάρχει ε, πρόβλημα παρόφεσης, αλλά υπάρχει και ένα ε, θέμα πιστοποίησης ε, ουσιαστικά και επιβεβαίωσης και βρισκόμαστε σε αυτή την ευρωϊκή κατάσταση γιατί αυτά τα σχέδια που σας ανέφερα πριν ε, που είχαν χρηματοδοτηθεί μέση χρηματοδότηση που αφαιρέθηκε ε, μείναν για ε, να περάσουν στον προγραμματισμό 2014-2020. Τα ξαναβλέπουμε τώρα, δηλαδή όσα είναι φυσικά ε, συμβατά με τη δική μας στρατηγική. Οι πληρωμές είναι μια σημαντική παράμετρο, το είπα αυτό στις ε, διαφάνειες, το είδαμε και στις διαφάνειες του Δενού Συναδέλφου, ε, δηλαδή είπα ότι πρέπει να σεβόμαστε τους κανόνες και να μην τους αφισβητούμε, όμως εδώ πρέπει να δούμε ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να εισαγάγουμε. Από την πλευρά μας λοιπόν, στην Ιταλία, εφαρμόζονται όλα αυτά τα μέτρα για να καταλάβουμε αν ε, τα σχέδια εξυπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες. Και ίσως η Ιταλία είναι η μόνη χώρα που έχει μια στρατηγική εξειδικεύσης για κάθε περιφέρεια και μια εθνική στρατηγική. Και αυτές ε, οι ε, στρατηγικές, τις περιοχές που σημειώνουν καθυστέρηση στην απορρόφηση, εισήχθησαν με προσπάθεια να υπάρχει διάλογος με την εταιρική σχέση και κατόπιν εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ήταν κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Η Σικελία έχει μία ε, πάρα πολύ αξιόλογη στρατηγική. Ήρθε λοιπόν σε επικοινωνία με πάνω από 60 ε, επιχειρήσεις, πανεπιστήμια κτλ. Όλα αυτά θα μας βοηθήσουν ε, όχι μόνο να προωθήσουμε τον προγραμματισμό, αλλά θα μπορέσουμε να δώσουμε και ένα καινοτόμο μήνυμα και ποιοτικό μήνυμα ε, και νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πλέον τόση καθυστέρηση. Σας δίνω λοιπόν ε, καλά νέα, δίχως να διασφαλίζουμε ότι έχουμε βγει από την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δοθεί σε αυτές τις περιοχές. Η δράση της ε, Task Force σίγουρα θα συνεχίσει. Όμως τώρα κάνουμε ένα διάλογο με τις διαχειριστικές αρχές, ε, τις αρχές πιστοποίησης και τις αρχές ελέγχου σε ένα πολύ πιο διαρθρωμένο πλαίσιο, γιατί έχουν υιοθετήσει μία μέθοδο και έχουν μάθει τα διδάγματα του παρελθόντος. Επιτέλους, κάποιο, κάποιες καλές ειδήσει. Έφτιαξε και ο καιρός πάνω στην ώρα, μια ωραία μέρα. Συνεχίζουμε με το πρόγραμμα και έχουμε τώρα τον κύριο Κάρλος Μέντες για να ακούσουμε την ακαδημαϊκή <clears throat> οπτική. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Γεια σας, ε, καλησπέρα σας. Κυρία Πρόεδρε, μέλη των άλλων θεσμικών οργάνων, θα ήθελα να πω δύο λόγια για ένα ερευνητικό πρόγραμμα, πρόγραμμα συγκριτικής έρευνας του, Ευρωπαϊκού, του Κέντρου Ευρωπαϊκών Πολιτικών για το θέμα της οικονομικής απορρόφησης. Ξέρω ότι έχουμε καθυστερήσει και γι' αυτό θα επικεντρωθώ στα βασικά σημεία. Υπάρχει πολλή βιβλιογραφία για την απορρόφηση, αλλά αυτά είναι παλαιότερα. Μελετώντας όλα αυτά, οι βασικοί παράγοντες είναι η ποιότητα της κυβέρνησης και των δικαιούχων ε, και επίσης ε, η ευρύτερη ποιότητα της ε, πολιτικής της κυβέρνησης θέματα και της πολιτικής της επιχειρηματικότητα, θέματα πολιτικής αστάθειας, θέματα εκλογών μπορεί να επιβραδύνουν την απορρόφηση, επίσης η κατάχρηση των ταμείων, η δομή, η θεσμική δομή, συγκεντρωτική, αποκεντρωμένη, επίσης τα κίνητρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κυρώσεις και βεβαίως η εκμάθηση. Παρά τις ε, περιορισμένες δυνατότητες, τα κράτη-μέλη, τα νέα κράτη-μέλη πήγαν καλύτερα όσον αφορά την δαπάνη και την συμμόρφωση κατά την πρώτη προγραμματική περίοδο. Όσον αφορά τις μελέτες αξιολόγησης η Γενική Διεύθυνση Ρέτζο ε, δημοσίευσε την εκ των υστέρων αξιολόγηση που έδειξε ότι το 2007-2013 ήταν βραδύτερη από ό,τι σε προηγούμενες περιόδους. Είναι ενδιαφέρον που το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο κατά την παρουσίαση του προηγουμένως είπε ότι οι δαπάνες ήταν συγκρίσιμες και στις δύο περιόδους. Δεν έχω καταλάβει γιατί το λέει αυτό. Ενδεχομένως να περιλαμβάνονται διαφορετικά ταμεία. Κάτι υπάρχει στα δεδομένα που θα πρέπει να το μελετήσουμε. Πάντως η εκ των υστέρων αξιολόγηση κατέληξε ότι η περίοδος μέχρι το 2013 ήταν βραδύτερη από ό,τι ε, νωρίτερα και επίσης ε, βραδύτερη από το 94-99. Η κρίση ήταν βασικός παράγων, αλλά αυτή αντιμετωπίστηκε με την ανταπόκριση Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, προπαταβολές, αλλαγές στα ποσοστά συγχρηματοδότησης, επίσης το ΠΑΠ οι αδυναμίες στα συστήματα επίδοσης, παράδοσης ήταν αιτίες δυσκολίες ε, στα, στις δυνατότητες των συστημάτων, οι δυσκολίες στην επιλογή των προγραμμάτων, αναφέρθηκαν προγράμματα στη Βουλγαρία, θέματα ε, στη Ρουμανία και στην Κροατία και θέματα επίσης ε, με τη διαχείριση των προσκλήσεων για πολύ ενδιαφέροντα, το, συνθ, το των κανονισμών και στο ευρωπαϊκό επίπεδο και στο ε, εσωτερικό των χωρών. Επίσης, μεγάλη κινητικότητα του προσωπικού, αυτό αναφέρθηκε στη Ρουμανία. Επίσης, η δυνατότητα δημιουργίας υποδομών, ε, μάθησης, η αποκέντρωση, ο κεντρικός συντονισμός, η απορρόφηση ε, δεξιοτήτων. Ακούσαμε για την Πολωνία και ακούσαμε και από άλλους συναδέλφους ότι υπήρχε ένα θέμα συντονισμού παλαιότερα. Εδώ βλέπετε τις διακυμάνσεις στο ε, ρυθμό και το χρόνο της, ε, ροή, της απορρόφησης ε, με την εξαίρεση της Κροατίας εντοπίζονται τέσσερις ομάδες εδώ από μια μελέτη κλεισίματος που έγινε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βλέπετε ότι ταξινομούνται οι διάφορες ομάδες κρατών μελών ανάλογα με τα επίπεδα Απορρόφηση το 2013 και ο ρυθμός μέχρι το 2016. Βλέπουμε διακυμάνσεις ανάμεσα στις χώρες. Το επίσημο κλείσιμο των προγραμμάτων και η μελέτη τους έδειξε ότι το κλείσιμο ήταν αποτελεσματικό όσον αφορά την υποβολή και την συμμόρφωση, αλλά δεν μελετήθηκε η ποιότητα των εγγράφων. Αυτό είναι μια εργασία που συνεχίζεται. Ο κύριος Πόπενς ανέφερε ότι οι εκθέσεις ε, ε, κλεισίματος θα εξακολουθήσουν να αξιολογούνται τους επόμενους μήνες οι πιέσεις ε, ε, δημοσιονομικής ε, απορρόφησης επηρεάστηκαν και επηρέασαν, αλλά αυτές αντιμετωπίστηκαν από διάφορες ευρωπαϊκές διατάξεις. Και για την περίοδο 2007-2013 ε, είδαμε ότι η αυστηρότητα του ελέγχου αυξήθηκε σε όλη τη διάρκεια της περίοδου και όχι μόνο στο τέλος. Επίσης ε, έγινε καλύτερη ε, υλοποίηση η συνεργασία μεταξύ ομοτήμων οδήγησε σε μια υποστήριξη προς τα κράτη-μέλη η υλοποίηση των ε, δημοσιονομικών εργαλείων και τα μεγάλα έργα ε, επηρέασαν το κλείσιμο, υπήρξαν καθυστερήσεις ε, γιατί καλύπτει μεγάλο ποσό της χρηματοδότησης. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία είχαν καθυστερήσεις, οι διάφορες αρχές δεν χρειάστηκε να, δεν μπορούσαν να ελέγχουν τα εργαλεία στη διάρκεια της φάσης υλοποίησης, αλλά κατά το κλείσιμο. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι το, η ποιότητα του κλεισίματος εξαρτάται κυρίως από την διοικητική δυνατότητα και την προσέγγιση της, ε, της κυβέρνησης και των αρχών. Η διαχείριση του κλεισίματος είναι δύσκολη και για τη διαχειριστική αρχή και για τις ελεγκτικές αρχές. Επίσης αυτό επιβαρύνεται έτσι περαιτέρω από τη μεγάλη κινητικότητα του ε, προσωπικού και από άλλους παράγοντες. Η έρευνά μας ε, στα πλαίσια του προγράμματος IQNet, που είναι ένα δίκτυο εθνικών και περιφερειακών αρχών, έδειξε ότι η εμπειρία της περίοδου 2014-2020 όσον αφορά την ζήτηση για προγράμματα ήταν καλή αλλά υπήρχαν δυσκολίες με πιο πρόσφατα και νέα και σύνθετα θέματα, θα επανέλθω σε αυτό. Επίσης, σαφής βελτίωση στην ποιότητα των αιτήσεων, πιο ε, απαιτητική η αξιολόγηση και επιλογή των προγραμμάτων, αυξήθηκε το ποσοστό των δεσμεύσεων οι περιορομές είναι πολύ περιορισμένες, κυρίως προκαταβολές τα πρώτα χρόνια και επίσης υπάρχει κάποια επιφύλαξη όσον αφορά τα αποτελέσματα, κυρίως όσον αφορά την επίτευξη των στόχων. Επανέρχομαι στο θέμα το βασικό θέμα, γιατί είναι σχετικά βραδίες οι πληρωμές, όπως επισήμανε και ο κύριος Πυρίνσκι, υπάρχει το θέμα της καθυστέρησης στην έναρξη του προγράμματος, οι καθυστερήσεις στο χρηματοοικονομικό πλαίσιο. Ο βασικός παράγων είναι οι καθυστερήσεις στη διαδικασία ορισμού. Αυτό αναφέρθηκε και από τις προηγούμενες παρουσιάσεις. Το 2015 μόνο το 1 τέταρτο των φορέων, των προγραμμάτων και των ενδιάμεσων φορέων είχαν οριστεί. Υπήρξαν σοβαρές καθυστερήσεις στο διάστημα αυτό για τον ορισμό των αρχών και τη δημιουργία των συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης. Αυτό είναι ένας ουσιαστικός παράγων που έχει σχέση και με τις νέες απαιτήσεις της περίοδου. Η αξιολόγηση συμμόρφωσης ε, ανατέθηκε στα κράτη-μέλη Επίσης έπρεπε να αντιμετωπιστούν νέες απαιτήσει, ε, κανονισμοί κατά της απάτης, αλλαγές στα ηλεκτρονικά συστήματα. Αυτό επηρέασε τις διαδικασίες ορισμού, οι οποίες ε, ολοκληρώθηκαν το 2016, ο τέλος του 2016. Επίση υπήρχαν και κάποια θέματα με την αλληπικάλυψη περιόδων. Δηλαδή, η ε, καθυστέρηση της απορρόφησης του 7 ως 13 είναι πλάκη με, την, το κλείσιμο και ε, ε, ε, έγινε μια προσπάθεια να γίνει πλήρης απορρόφηση των προηγούμενων κονδυλίων ενώ πριν αρχίσουν τα επόμενα. Επίσης υπάρχει ο στόχος της οικονομίας με χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Υπάρχουν πολλοί νέοι δικαιούχοι εδώ, επισέρχονται νέοι παράγοντες και νέα μέσα, νέα ε, εδαφικά εργαλεία, ε, βιώσιμη αστική ανάπτυξη και επίσης ολοκληρωμένες ε, χωροταξικές επενδύσεις που καθυστέρησαν την εφαρμογή χρηματοοικονομικά μέσα που άρχισαν να ξεκινήσουν παρότι εκεί έχουν γίνει βελτιώσεις. Ας πούμε, σχεδιασμός της εκ των προτέρων αξιολόγησης είναι κάτι που χρειάζεται σε αυτή την περίοδο και τουλάχιστον αυτό βοηθά να εντοπιστούν να εντοπιστεί μια πιο εξορθολογισμένη βάση για τα μέσα που στο μέλλον θα βοηθήσουν την απορρόφηση η αλληλουχία των διαφόρων μεριδίων της χρηματοδότησης, ότι ώστε οι καταβολές να γίνονται αφού έχουν δοθεί τα χρήματα στους δικαιούχους. Όλα αυτά θα βοηθήσουν τα χρηματοοικονομικά εργαλεία, αλλά υπήρχε μια επιβράδυνση. Επίσης υπήρξε και η πίεση της χρηματοδότησης λόγω της δημοσιονομικής εξυγένσης σε κάποιες περιπτώσεις. Επίσης υπήρχε διακυμάνσεις ε, της, ε, του συναλλαγματικές διακυμάνσεις ανάλογα με τις χώρες και οι ε, επιστροφές από τα χρηματοοικονομικά εργαλεία μπορούν να επηρεάσουν το σχεδιασμό. Θέματα συμμόρφωσης, η εκ των προτέρων ερεσιμότητα ήταν ένα νέο στοιχείο αποτέλεσε σε μερικέ περιπτώσεις μεγάλο διοικητικό βάρος και χρειάστηκαν και προγράμματα δράσης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο επίσης υπήρχαν θέματα συγκεκριμένα ε, σε σχέση με το Brexit που σταμάτησε πολλά προγράμματα και πολλές δαπάνες τα βασικά μέτρα για την υποστήριξη της, ε, την ενίσχυση της απορρόφησης είναι τα αριθμιστικά, αναθεώρηση της εσωτερικής νομοθεσίας, δηλαδή εξορθολογισμός ή απλούστευση των διαδικασιών προμηθειών, ε, και σε, ε, σε, σε επίπεδο προγραμμάτων, η αναθεώρηση των προγραμμάτων, η ανακατανομή των κονδυλίων ανάλογα με τι προτεραιότητε, σε επίπεδο έργου, ο συντονισμός και η, προτεραιότητα διαφόρων προσκλήσεων ε, ενδιαφέροντος από τα ευρωπαϊκά διορθωτικά ταμεία και ταμεία επενδύσεων, τα μπόνους τη χρηματοδότηση, τα τριγικά προγράμματα και επίση ενημερωτικέ εκδηλώσει που έγιναν για του δικαιούχου. Όσον αφορά, επειδή μάλλον μου μίλησαν να μιλήσω για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Η συζήτηση για την αναθεώρηση έχει μόλις ξεκινήσει. Η Κομισιόν πρόκειται τώρα να δημοσιεύσει την έκθεση συνοχής αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει πολλαπλές κρίσεις. Χρηματοοικονομική κρίση, οικονομική κρίση, κρίση μετανάστευσης, με τις επιπτώσεις που έχει αυτή τη, στην ανισότητα. Ακούσαμε ότι το, ο μηχανισμός σύγκλησης έχει καθυστερεί. Ένα πολύ δύσκολο πλαίσιο για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής ενοχής. Μια πρόσφατη μελέτη που παρουσιάστηκε στο Φόρουμ Συνοχής ε, από τον καθηγητή Τζον Μπάκλεϊ, και μια σειρά άλλους καθηγητές υποστηρίζει ότι αυτό το οποίο χρειάζεται είναι μια ισχυρή ευρωπαϊκή πολιτική δέσμευση ε, ε, σε σχέση με την πολιτική πραγματικότητα, όχι μόνο ανάπτυξη εν γέννη, αλλά όλες οι περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η παγκοσμιοποίηση. Σε συνδυασμό με ταχύτερη και ισχυρότερη έμφαση στην χωροταξική διάσταση της πολιτικής συνοχής. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για την ευθυγράμμιση της πολιτικής συνοχής με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούσαμε προηγουμένως για την ευθυγράμμιση της, του θεματολογίου της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης γίναν προτάσεις, αυτή είναι η σχέση με την πολιτική συνοχή, τη δυνατότητα να προχωρήσουμε προς τα εκεί. Επίσης, η ευθυγράμμιση με τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου υποτηρίζεται εδώ ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο πρέπει να λάβει περισσότερο υπόψη του την χωροταξική διάσταση της πολιτικής συνοχής, ώστε η πολιτική συνοχή να μην θεωρείται μόνο όχημα για να φτάσουμε ε, στους στόχους του Ευρώπης 2020 για την οικονομική διακυβέρνηση, αλλά ε, στην πορεία ε, να λάβει υπόψη της τη συνοχή. Η συνοχή θεωρείται ότι εμπίπτει σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένες και της οικονομικής πολιτικής που αποτελεί και υποχρέωση συνθήκη, από τη συνθήκη. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, οι επιδόσεις και τα αποτελέσματα ποικίλουν. Υπονομεύονται από τις αδυναμίες στο θεσμικό πλαίσιο, την πολιτικοποίηση, ε, τη διοικητική δυνατότητα Υπάρχει και ένα θέμα που συζητείται σχετικά με τις εκ των που ε, υπάρχουν παρεμβάσεις που ισχυρίζονται ότι είναι πολύ χρήσιμες στην Ρουμανία και την Ιταλία γιατί ενισχύουν τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική ε, υλοποίηση. Ο κύριος Πόπενς υπογράμμισε τη σημασία του να υπάρχουν στρατηγικές για την διευκόλυνση της χρηματοοικονομικής ε, απορρόφησης, όμως εδώ η βασική στόχη είναι πόσο νόημα έχουν, πόσο χρήσιμα είναι τα διαρθρωτικά ταμεία στο περιφερειακό πλαίσιο. Ένα ζήτημα είναι να προσπαθήσουν να περιοριστούν οι ο αριθμός των αιρεσιμοτήτων στο μέλλον ώστε οι αρχές των κρατών, οι αρχές των κρατών μελών έχουν επικρίνει την έλλειψη συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τον επανέλεγχο των, της αιρεσιμότητας από τις διάφορες γενικές διευθύνσεις. Ένα άλλο ζήτημα αφορά η παροχή, την παροχή κινήτρων σε σχέση με την αιρεσιμότητα. Δεν είναι μόνο θέμα ενός καταλόγου που πρέπει να ε, ολοκληρωθεί, αλλά πρέπει τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες να έχουν κίνητρα για να αναλάβουν αυτούς τους όρους που τους τίθενται. Υπάρχει ένα θέμα που αφορά ε, ε, περισσότερο, περισσότερη έμφαση στην δημιουργία διοικητικής δυνατότητας και αυτό έχει σχέση με συστήματα παράδοσης αν θέλετε με συστήματα που βοηθούν την αποτελεσματικότητα οι πληρωμές που στηρίζονται στις, στην απόδοση ή στους στόχους αυτό από μόνο του όμως θα απαιτούσε τον υπολογισμό ενός ε, σταθερού τυποποιημένου κόστους. Τώρα, ένα άλλο θέμα είναι ένα ευρύτερο ε, αφήγημα δημόσιο και από τα μέσα ενημέρωσης. Είναι αρνητικό. Προσπαθούμε τώρα να φέρουμε την πολιτική συνοχή πιο κοντά στους πολίτες, να γίνει πιο θετικό το αφήγημα. Η συζήτηση είναι μάλλον καταστροφική σε σχέση με τον ε, ε, προϋπολογισμό και τις περιοδικές ε, μεταρρυθμίσεις του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Πολλοί λένε ότι είναι τεράστιος ο προπολογισμό, είναι δαπανηρός, ότι γίνονται σπατάλες, ότι ε, πρέπει να αναγνωριστεί η αλληλεγγύη. Και μοιάζει ότι υπάρχει μια έμφαση στο ε, εσωτερικό της Ένωσης σχετικά με την συμμόρφωση. Η διαδικασία απαλλαγής του προπολογισμού έχει μια αρνητική ε, έννοια και θεωρείται ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση βρίθη απατών και ελάχιστα ε, αναγνωρίζονται οι ευρωπαϊκές δαπάνες. Η χρηματοδότηση είναι μόνο μέρος των επενδυτικών έργων. Πολύ συχνά η διαφήμιση θεωρείται ότι είναι η προπαγάνδα. Όλα αυτά είναι αρνητικά και ο συνολικός τόνος από τα μέσα ενημέρωσης και την κοινή γνώμη είναι μάλλον αρνητικός. Δεν είναι πάντοτε έτσι, αλλά το επιχείρημα είναι ότι μια ε, ισχυρότερη και πιο αποτελεσματική επικοινωνία ε, ε, είναι απαραίτητη. Χρειάζεται να υπάρχει μεγαλύτερη επαφή με τους πολίτες για να φύγουμε από τα θέματα της απορρόφησης και της συμμόρφωσης και να επικεντρωθούμε στα επιτεύγματα και στο πώς επηρεάζεται η καθημερινή ζωή των πολιτών. Επίσης έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για την ευελιξία, την, ώστε να ανταποκρινθούμε στις δυσκολίες αυτό αφορά κυρίως το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Υπάρχουν δυνα... διάφορες δυνατότητες ώστε να διευκολυνθεί και η απορρόφηση και η αναθεωρήση των του προγραμμάτων με βάση την παλαιότερη εμπειρία, τα αποθεματικά των προγραμμάτων, τα ε, αποθεματικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούσαμε ότι η ιστορία της πολιτικής συνοχής ήταν μια μεγάλη πρόκληση στον τομέα της ε, διακυβέρνησης λόγω του σύνθετου χαρακτήρα των κανονισμών, τα διαφορετικά επίπεδα ε, διοίκησης και η Ιταλική παρουσίαση είχε μια ε, παρόμοια διαφάνεια για τις διαφορετικές διατάξεις που εμφανίστηκαν σύντο χρόνο. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν και επηρεάζουν την απορρόφηση σε κάθε νέα περίοδο. Υπάρχει και η δυσκολία των ελέγχων και ο φαύλος κύκλος των ελέγχων όπου οι υπερβολές επικρίνονται από τις δημοσιονομικές αρχές, ε, το ελεγκτικό συνέδριο. Αυτό οδηγεί σε νέες ρυθμιστικές απαιτήσεις που προκαλούν αβεβαιότητα. Ακούσαμε τον κύριο Γκρέξον ε, που μας είπε ότι αυτό ε, βρίσκεται πίσω από τα αιτήματα των κρατών μελών για νέες ερμηνείες, καθοδήγηση που οδηγεί σε νέες διαδικασίες, νέους κινδύνους και πιθανώς περισσότερα σφάλματα. Αυτό που χρειάζεται, κυρίως κατά την άποψη των διαχειριστικών αρχών με τις οποίες συνομιλήσαμε, είναι η απλούστευση των κανόνων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητη να υπάρχει, απαραίτητο να υπάρχει μόνο ένα σύνολο κανόνων για τα κράτη-μέλη που έχουν μικρά ποσά, αυτό θεωρείται ανεπαρκές. Ζητάνε μια πιο βαθιά αλλαγή στη... στον τρόπο διαχείρισης που έχει σχέση και με την αποδοτικότητα της απορρόφησης, την αποδοτικότητα των δαπανών και όχι αυτή καθε αυτή την απορρόφηση. Γιατί το κόστος, το διοικητικό βάρος έχει σχέση που συνδυάζεται με την υλοποίηση των προγράμμων θεωρείται πάρα πολύ ψηλό με που, σε χώρες που τα κονδύλια είναι χαμηλά. Και αυτό μπορεί να στηρίζεται στις αρχές του κινδύνου ή στην προσέγγιση με βάση το αποτέλεσμα, τους εθνικούς κανόνες υλοποίησης, μεγαλύτερη ε, σχέση με εθνικούς ελέγχους και επίσης τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. Πιθανά κριτήρια διαφοροποίησης θα μπορούσαν να είναι. Το επίπεδο χρηματοδότησης, η κλίμακα δηλαδή των κονδυλίων, το επίπεδο ευρωπαϊκού, ευρωπαϊκής ε, συγχρηματοδότησης και το ποσοστό των επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ ή ως προς το, ε, τις δημόσιες επενδύσεις. Άλλα κριτήρια μπορούν να, έχουν, να λάβουν υπόψη τις, το ποσο, τις επιδόσεις, την υλοποίηση, την απορρόφηση, τις παρατυπίες ή πάλι την διοικητική δυνατότητα. Δεν υπάρχουν διοικητικοί δείκτες γι' αυτό, αλλά έχουν γίνει κάποιες έρευνες για την ποιότητα της κυβέρνησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Εν κατακλείδη, όσον αφορά το τι θα συζητηθεί στο μέλλον. Η ενίσχυση της χωροταξικής διάστασης μοιάζει απαραίτητη για να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες, κυρίως όσον αφορά λόγω της κρίσης και τη έλλειψη διαφοροποίησης, μια μεγαλύτερη ευθυγράμμιση της οικονομικής διακυβέρνησης και της πολιτικής συνοχής, η ενίσχυση και η προσαρμογή των, της εκ των προτέρων ερεσιμότητας, πιο αποτελεσματική επικοινωνία, μια αλλαγή στο φύγημα, η ευελισία για στη, ώστε να υπάρξει προσαρμογή στη νέα, σε νέες κρίσεις, σε νέα ζητήματα και ευελιξία για την μεταρρύθμιση των προγραμμάτων στο εσωτερικό τους και απλούστευση έτσι ώστε να υπάρχει μια περισσότερο διαφοροποιημένη προσέγγιση στην ε, διαχείριση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία απαλλαγή όμω, ε, δημιουργήθηκαν κάποιε απορίε. Και τα περί απάτης. Έχετε διαβάσει, μάλλον δεν έχετε διαβάσει τι εκθέσει μα περί αλλαγής. Νομίζω ότι έχουν βελτιωθεί πολύ αυτές οι εκθέσεις και νομίζω ότι θα πρέπει να τα δείτε κάπως διαφορετικά. Δεν κατάλαβα ακριβώ τι εννοείται με την territorial dimension ακριβώς, την χωροταξική αυτή διάσταση. Κάποιοι όταν βλέπουν ότι υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια μπορεί να το θεωρούν καλό, αλλά το πρόβλημα είναι η επικοινωνία. Στα διαρθωτικά ταμεία έχουμε 400 δις, τα οποία τα κατανέμουμε μέσα στην επταετία. Λίγο λιγότερα, λίγο περισσότερο. Είναι δυνατόν να φανταστεί κανείς ότι δεν υπάρχουν αποτελέσματα με αυτά τα κονδύλια. Απλά εμείς αυτό που μας επασχολεί είναι να βελτιώνονται τα αποτελέσματα υπάρχουν κάποιοι που παίρνουν πολλά κονδύλια για πολύ καιρό και δυστυχώς ε, κοιτάω ε, προς την Ιταλία. Αλλά ε, βλέπουμε οι επιδόσεις να μην είναι τόσο καλές. Και το ελεγκτικό συνέδριο, όπως κάθε χρόνο, μας ε, στέλνει 35 με 36 ειδικές εκθέσεις, τις οποίες μελετάμε. Και πρέπει να σας πω ότι και η γάμα δέλτα Ρέγγιο δεν τα παρουσιάζει τα πράγματα σωστά. Έχουμε κάνει πολύ σημαντικά πράγματα. Παραδείγματος χάρη στην Πολωνία έγιναν πολύ καλά με τα χρήματα αυτά. Σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των μέσων, τα χρήματα δόθηκαν αλλά ο Πολωνός πολίτης δεν ε, είχε κάποια συμμετοχή, δεν είχε ενημέρωση. Αυτό είναι το πρόβλημα, πιστεύω. Πώς θα εξηγήσουμε ότι εσείς για την ίδια απόδοση δεν για παράδειγμα, πρέπει να πληρώσετε από την τσέπη σας, ενώ άλλοι υποφελούνται ε, χωρίς να δαπανίσουν ούτε ένα σέντα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το συζητήσουμε και θα το κάνουμε και στο μέλλον. Έχω και κάποιες ερωτήσεις σε σχέση με την εμπειρία σας για τη διοικητική ικανότητα. Υπάρχει χρήμα, υπάρχουν μέτρα που μπορούμε να προωθήσουμε. Πάντα βλέπουμε όμως ότι είναι δύσκολο να αξιολογούμε την δίκηση, αλλά μετά αν υπάρχουν προβλήματα πηγαίνουν οι άνθρωποι σε κάποιες ε, ειδικέ εταιρείε ε, οικονομικού ελέγχου ή σε άλλους συμβούλους. Δεν είναι λοιπόν τόσο απλά τα πράγματα. Η κατηγορία μας, αν θέλετε, προς την Κομισιόν είναι ότι σε κάποια κράτη-μέλη θα μπορούσαν να είναι πολύ καλύτερε οι επιδόσει αν ήταν σαφέ από την αρχή. Πώ θέλουν να πετύχουν αυτά τα αποτελέσματα, διότι έχουν ε, εγκριθεί κάποια προγράμματα τα οποία μετά κανένα δεν τα θεωρεί καλά. Και υπάρχουν άλλα πολύ καλά προγράμματα. Ή άλλα τα οποία είναι μόνο κατά το ίμιση επιτυχημένα. Τα έχουμε δει και πρέπει να μας απασχολήσει και αυτό το θέμα και πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τέτοια φαινόμενα. Αυτά ήταν η δική μου παρέμβαση και θέλω να δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Πυρίνσκι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Ήταν πολύ ευρία η παρουσίαση που αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα του, περι... του πλαισίου και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση. που έχουν περιπλακεί ακόμη περισσότερο με το παρελθόν. Έχω μία ερώτηση προς τον κύριο Μέντες που μας έδειξε ένα γράφημα με τέσσερις ομάδες χωρών με διαφορετικά προφίλ απορρόφησης πρόωρη, με, μεσαία, καστερμένη, πολύ καστερμένη. Πώς τη μετράμε την ταχύτητα της απορρόφησης. Στις χώρες εντός αγικών είναι και η Δανία. Και ο κ. Δανία το είπε στην παρουσίασή του, ότι του έχει ασκηθεί κριτική για καστερημένη απορρόφηση. αλλά μιλούσε για δεσμεύσεις. Και μια άλλη πτυχή που ανέφερε και ο παρουσιαστής αυτής της μελέτης είπε ότι υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις μεταξύ των πορισμάτων του ελεγκτικού. Ότι περίπου ίδια ήταν τα ποσοστά πορισμής προηγούμενες περίοδους. Και αυτό έρθει σε διαστολή με τη δική του δήλωση ότι υπήρξε βελτίωση στις δύο τελευταίες σε σχέση με την προηγούμενη. Εμείς εδώ θέλουμε να αξιολογήσουμε σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων ως προς την απορρόφηση. Είπατε ότι υπάρχει μια συνέχεια μεταξύ τριών ομάδων ζητημάτων που είναι η συμμόρφωση, η απορρόφηση και τα αποτελέσματα. Αν κατάλαβα καλά τουλάχιστον. Ποιο είναι ο σχετισμό μεταξύ των τριών πτυχών και πώ μπορούμε αντί τη μία να την φέρνουμε αντιμέτωπη με την άλλη, τι τις να τι εναρμονίσουμε μεταξύ του, Κυρία Σέντερ. Ευχαριστώ. Και εγώ είχα τον ίδιο προβληματισμό με τον κύριο Πυρίνσκι και καθώς έχω την τιμή να κάθομαι εδώ δίπλα στον κύριο Γεγίρσαν μπορούσα να του κάνω αυτή την ερώτηση γιατί ακριβώς ε, για μένα μετά την παρουσίαση ήταν κάπως παράξενο να παρουσιάζονται η Δανία σαν καθυστερημένη στην απορρόφηση, ενώ εμείς να είμαστε στη μεσαία θέση. Ίσως αυτό είναι κάτι που δεν το συζητήσαμε, αλλά να σχετίζεται με το πώς μετρούνται και τα αποτελέσματα σε έναν πολυετή προϋπολογισμό και που όλοι ξέρουν ότι υπάρχουν αυτά χρόνια και υπάρχει και ο κανόνα νη 1, ή 2, νη 3 για την εφαρμογή. Τελικά το φωτοφίνη ε, που κάνει το ελεγκτικό συνέδριο, για να μην ε, πούμε εμεί, είναι ετήσιο. 2013. Ε, Στην αρχή θα έγινε ένα φωτοφίνης της απορρόφησης της Δανίας. Ε, βρισκόμαστε στο 48% πριν Οσχαρή, που το θα σκούσαμε κριτική. Ενώ αν πάμε στο 2015 βλέπουμε ότι είναι στο 100%. Εγώ συγγνώμη, πρέπει να φύγω, όμως ε, μου το είπε ο κύριος ε, Γκρέγκερσεν το μυστικό. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα άλλο τμήμα της πολύπλοκης δουλειάς μας. Δηλαδή αξιολογούμε και μετρούμε τήσιους προϋπολογισμούς ε, σαν να βρισκόμαστε σε εθνικό επίπεδο, όμως ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε πολιετής προϋπολογισμούς ε, και φυσικά αυτό επιφέρει πολυπλοκότητα. Έτσι λοιπόν το φωτοφινής δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντικατοπτρίσουμε την πραγματικότητα. Εγώ συγγνώμη που πρέπει να φύγω, αλλά σίγουρα ο κύριος Πυρίνς και ο συνάδελφος ε, θα μου πει αν θα προσθέσετε κάτι σε αυτό το μυστικό. Ο κύριος Μέντες. Ευχαριστώ. Το πρώτο θέμα όσον αφορά την απαλλαγή αφορά περισσότερο το πώς γίνεται αντιληπτό το θέμα αυτό. Η, η απαλλαγή είναι σωστή, είναι απαραίτητη, βρίσκονται σφάλματα και πρέπει να αναφέρονται. Σημασία έχει όταν αυτό το αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης, τότε η τάση είναι να παρουσιάζεται με αρνητική, από αρνητική σκοπιά. Το δεύτερο θέμα αφορά τη χωροταξική διάσταση. Ε, αναφέρθηκα σε μια έκθεση που ε, αφορούσε την πολιτική συνοχής 4.0 και έδειχνε ότι το γεγονός ότι συντο χρόνο η πολιτική συνοχής απέκτησε μια τομεακή ή θεματική, λογική, θεματικούς στόχους που συχνά οδηγούν σε πιο περιορισμένη σκέψη σε επίπεδο περιφερειακό ή υποπεριφερειακό όσον αφορά το σχεδιασμό των προγραμμάτων. Βλέπουμε δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις ότι δεν ε, τα, ανταποκρίνονται στα προγράμματά τους τις ανάγκες της περιφέρειας αυτές καθεαυτές, αλλά ξεκινούν από τις θεματικούς στόχους και προγραμματίζουν τη χρηματοδότηση σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες τους. Αυτή είναι μία από τις πλευρές της λογικής που περιέγραψα. Είπα επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο που και αυτό έχει μια προσέγγιση περισσότερο ε, τομεακή, πιο εθνική, δεν λαμβάνει κατά ανάγκη υπόψη του τις διαφορές ανάμεσα στις διάφορες περιφέρειες. Αυτό, η αφορά, αυτό, είναι, αυτό ήθελα να πω όσον αφορά τη χωριατεξική διάσταση. Η γενική κατεύθυνση είναι ότι στο διάστημα αυτό έχει επέλθει αλλαγή. Οι λογικές παρέμβασεις είναι πολύ πιο σαφείς στα προγράμματα από ό,τι ήταν στο παρελθόν ο κύριος Γκρέγκρτσον έδωσε ένα παράδειγμα σε επίπεδο έργου, αλλά σε επίπεδο προγράμματος, ο σχεδιασμός του προγράμματος, με βάση τους διάφορους δείκτες, η λογική των παρεμβάσεων, οι προτεραιότητες των επενδύσεων κλπ. έχουν βελτιωθεί σημαντικά στην περίοδο αυτή. Το είπε και ο κύριος Πόπενς. Το θέμα είναι ότι θα δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις όσον αφορά την επίτευξη των αποτελεσμάτων. Υπάρχει η άσκηση για το πλαίσιο επιδόσεων. Μερικές φορές ε, υπάρχουν ανησυχίε για την επίτευξη των ε, γενικών ε, στόχων επίδοσης άσχετα από το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αυτά είναι αυτά που πρέπει να παρακολουθήσει κανείς στη διάρκεια του χρόνου. Τέλος, διαφορές στο ρυθμό και στο χρόνο. Ξεκίνησε, ε, κυκλοφόρησε η έκθεση στα μέλη. Ε, δεν ε, έφτιαξα εγώ τα, τα γραφήματα για τα ποσοστά απορρόφησης. Ξέρω όμως ότι ποια είναι τα δεδομένα στην πλατφόρμα της Κομισιόν και έγινε σύγκριση ε, των δεδομένων του 13 με το 16. Δεν ξέρω για ποιο λόγο διαφέρουν τα ε, δεδομένα που προέρχονται από άλλες πηγές. Ενδεχομένως να περιλαμβάνονται προκαταβολές που πρέπει να ε, περιλαμβάνονται, δεδομένου ότι μερικές φορές αναφέρεται επίπεδο 95%. Οι επιδόσεις της Δανίας συγκεκριμένα, εγώ θεωρώ, με βάση το πώ είναι οργανωμένο αυτό, με βάση το ποσοστό απορρόφησης το 2013, θεωρείται καθυστέρηση στην απορρόφηση. Αυτό όμως δεν είναι κατά ανάγκη αρνητική παρατήρηση. Αφορά το προφίλ. Ίσως η Δανία να έφτιαξε ένα προφίλ που θα, έχει αυτή, που θα είναι τέτοιο, που θα έχει αυτή την εικόνα. Δεν είναι κατά ανάγκη κακό να θεωρείται κανείς, ε, να έχει κανείς καθυστέρηση στην απορρόφηση. Η μεγάλη καθυστέρηση είναι ανησυχητική. Γιατί έτσι δια, ε, ε, χάνονται οι επενδύσεις. Αυτά. Σε αυτό συμφωνούμε. Έχετε κάτι να πείτε, θέλετε να αντιδράσετε. If Λοιπόν, θέλετε να σας αποκαλύψω κάποια από τα μυστικά που είπα στην κυρία Γιαλασέντερ. Είναι αλήθεια ότι το αρχικό μου σχόλιο είναι όταν ε, συγκρίνεις τα ποσοστά παρόφηση. Είναι σημαντικό να κατανοήσεις ότι υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ της δέσμευσης των σκονδυλίων και δηλαδή της ανάληψης των υποχρεώσεων και της συγγραφής των συμβολέων, των πληρωμών δηλαδή. Ε, και πρέπει να γίνει η μέτρηση σε αυτή την κατεύθυνση. Από την περίπτωση της Δανίας, και αυτό το λέω χωρίς να το έχω προβλέψει, όταν ξεκινήσαμε την περίοδο 7-13, πήγαμε σε ένα δημαρχείο και γράψαμε την πολιτική μεταρρύθμιση ε, στη Δανία. Και εγώ ανέφερα ότι έπρεπε ουσιαστικά να ρηχτούν στη δουλειά και από 14 ε, κομιτείες θα έπρεπε να έχουν 5 ε, και από τις 200 δήμους θα έπρεπε να πάνε στους 98. Έτσι λοιπόν ε, το 2006 είχαμε αυτή την κατάσταση και αυτό μπορεί να μας καθυστέρησε, δεν το αρνούμε. Κάτι άλλο, όταν ξεκινάς μια νέα προγραμματική περίοδο, και αυτό ισχύει για τους περισσότερους, η εμπειρία που έχουμε είναι το εξή. Ένα νέο πρόγραμμα είναι σαν να φορά ένα νέο γάντι, δηλαδή σε στενεύει από αυτό που είχε πριν, γιατί θα συνηθίσει το άλλο γάντι, τώρα έχει ένα καινούριο γάντι και σε σφίγγει. νομίζω ότι το ίδιο βιώσαμε και εμείς όταν περάσαμε από τα παλιά προγράμματα που είχαμε σε προγράμματα εθνικής εμβέλειας. Αυτό μπορεί να μας καθυστέρησε κάπως. Όμως ήταν ουσιαστικά υπολεπτομερή έλεγχο και μελέτη στην Επιτροπή Παρακολούθησης και με τους desk officers της Κομισιόν και στις περιφερειακές γραμματείες. Εμείς ε, πολύ προσεκτικά χρησιμοποίησαμε τον κανόνα μη 2 και η εισαγωγή του κανόνα αυτού έχει μια συγκεκριμένη έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό. Για κάθε σύμβαση ε, είχαμε 1,5 χρόνο για να υποβάλουμε την έκθεση στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Αγκρό, ευχαριστώ. Ένα πολύ γρήγορο σχολείο. Ήταν ε, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση. Ο κοινοτικό ε, προπολογισμό και προπολογισμό ε, για την συνοχή αξιολογεί κατά νέμι τον ίδιο τρόπο τα ποσοστά για τα 7 ή για τα 10 χρόνια. Δηλαδή, η εμπειρία ξέρουμε ότι δεν μπορεί να είναι ίδια στην έναρξη. Πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε πάρα πολύ στην απορρόφηση. Γιατί αυτό που μετράει για το που, που κατευθύνεται η καμπύλη και για τη διαδρομή της, ε, αυτό μέτρα είναι στον νήσιν 2, δηλαδή να μην χάσουμε τους πόρους που έχουν δρομολογηθεί ποιο κάποιες επενδύσεις στο κράτος μέλος και να φτάσουμε στην πλήρη απορρόφηση. Πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε πάρα πολύ σε αυτό το θέμα, στο πώς δηλαδή μας λέει η εμπειρία ότι η κεντρική περίοδος ε, ξεκινά κάπως αργότερα, δηλαδή όταν γίνονται οι πληρωμές επιτόπου. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά όλους. Και για να κλείσει ο κύριος ο ηγητής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχω την εντύπωση ως καταληκτική παρέμβαση. Θα μπορούσα να πω πολλά, αλλά δεν θέλω να είμαι διεξοδικός και να απαντήσω όλα τα σχόλια. Απλά να συνοψίσω τα βασικά συμπεράσματα. Το πρώτο. Ποια είναι η λογική της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι συνοχή θα πει οικονομική, κοινωνική, εδαφική συνοχή. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν με μια ένωση και αγορά που θα λειτουργούν εύρυθμα. Σε ό,τι την επόμενη περίοδο προγραμματισμού θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε ακριβώς τον τρόπο τον οποίο εννοούμε την πολιτική αυτήν συνοχής και την έννοια της συνοχής για τα επόμενα βήματα και στο σχεδιασμό. Και το δεύτερο συμπέρασμα έχει να κάνει με την έννοια της απορρόφησης. Πώς τον ταχυριζόμαστε το δίκτυ αυτό που τον μετράμε καλύτερα με τα δαπανηθέντα ποσά. Τεράστιος αριθμός διαφορετικών παραγόντων αντικατοπτρίζονται. Οι κανόνες, δημοσιονομικά ζητήματα, διοικητική ικανότητα, χρονοδιάγραμμα, περιφερειακή διοίκηση. η απορρόφηση θα πρέπει να είναι ένα συναγερμός αν θέλετε που θα μας ε, εντοπίζει από πρόωρο στάδιο αν κάτι δεν λειτουργεί καλά ώστε να παίρνουμε τα μέτρα μας. Νομίζω το είπε και ο κύριος από το ελεγκτικό συνέδριο. Δηλαδή να υποβάλουμε αναφορές και να αντιδρούμε γρήγορα σε ό,τι το πλαίσιο. Έχουμε τη λειτουργία, τους κανόνες, τον προπολογισμό και έχουμε και τον προγραμματισμό σε αυτό το πλαίσιο. Και πάλι στο τέλος θα υπάρξει βιασύνη. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το Omnibus, ε, ούτε και με το πολιετές που είναι στον αέρα για όλους τους λόγους που ξέρουμε. Άρα είναι προφανές ότι θα πρέπει εδώ να αντιληφθούμε ότι έχουμε μία περίοδο που χαρακτηρίζεται από κρίση και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με πάρα πολύ καλή προετοιμασία γιατί δεν ακούσαμε τι κάνουν ότι δουλεύουν δύο χρόνια πριν την περίοδο και μετά προσπαθούν να προσαρμοστούν. Η Κομισιόν μας είπε ότι κάτι αντίστοιχο κάνουν. Έκαναν μάλλον πριν αρχίσει αυτή η περίοδος. Και φάνουμε στην διαπραγμάτευση και την έγκριση των προγραμμάτων που υποβάλλονται και εδώ πρέπει να επανέλθουμε στη λογική της συνοχής και τι θέλουμε να πετύχουμε. Θέλουμε μια πλήρη συνοχή. Και εδώ πρέπει να βρούμε, κυρία Πρόεδρε, την ισορροπία. Πόσο εξονοχιστικά θα ελέγχουμε την ποιότητα του κάθε ε, έργου και το πώς λειτουργεί κάθε αρχή, αφενός και τις δυναμικές που πρέπει να υπάρχει για να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Πράγματι υπάρχει και το θέμα των καθυστερήσεων στους ορισμούς, στους διορισμούς. Το είπε ο κύριος Μέντης. Αλλά μέχρι στιγμής πράγματι υπάρχει πρόβλημα. 16,8% των διχειριστικών αρχών δεν έχουν οριστεί. Υπάρχει ένας κίνδυνος, πραγματικός κίνδυνος για 95 επιχειρησιακά προγράμματα που θα περιοριστούν λόγω αυτόματης αποδέσμευσης αν δεν ληφθούν έκτακτα μέτρα για να μπορέσουν να ορίσουν τις διαχειριστικές αρχές στα κρατημέλη και να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα κονδύλια αυτά. Το να γραφούν δεν είναι αρκετό και είναι ανησυχητικό αυτό το φαινόμενο. Υπάρχει επίσης αυτό νέο πλαίσιο για τις σχέσεις πολιτικής συνοχής, επενδυτικού ταμείου, ε, διαρθρωτικών ταμείων με το blending των χρηματοδοτικών μέσων ταμείωσης κτλ. Νέες εξελίξεις ε, που συνιστούν όμως μια μεγάλη πρόκληση και πρέπει να υπάρξει προετοιμασία στην πράξη. Για να ολοκληρώσω, επανέρχομαι σε αυτό που προσπαθώ να σας πω από την αρχή. Ότι δηλαδή η Κομισιόν πρέπει να δώσει μεγάλη όθηση και έμφαση σε όλες αυτές τις πολύ μεγάλες προκλήσεις από την ενολογική σύλληψη της πολιτικής συνοχής μέχρι την εφαρμογή της. Το άρθρο 58 που περιλαμβάνει πολλά μέτρα τεχνικής ε, φύσεως που πρέπει να λάβει η Κομισιόν με δική της πρωτοβουλία για να αξιόλογηση και την εκτίμηση των προγραμμάτων και έργων. και να λάβει υπόψη και την έκθεση συνοχής κτλ. λοιπά. Ο κ. Πόπεν, στη δεύτερη ή τρίτη παρέμβασή του, to be a bit more attentive to the expectations <laughs> were. Ε, δεν νομίζω ότι πολύ κατάλαβε τι του ζητάμε, αλλά τέλος πάντων ναι, μας είπε να συνεργαστούμε, αλλά ναι, να συνεργαστούμε, αλλά να είμαστε σοβαροί. Να θέσουμε επιτάπητο στις προκλήσεις και τα πραγματικά στοιχεία. Πολύ χρήσιμη μπορούσε να είναι αυτή όλη η άσκηση, αλλά εάν λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά που μάθαμε σήμερα και αν είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε πάρα πολύ εντατικά με, με των προκλήσεων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. πρώτα πρώτος ευχαριστώ πολύ όλους τους συμμετέχοντες και το ελεκτικό συνέδριο θέλω να ευχαριστήσω. Αύριο το πρωί θα ασχοληθώ με την Ελλάδα. Θα είναι και γενικός διευθυντής Λεμέτρα. σε σχέση με το πρόβλημα ε, του κλεισίματος για την, του, του πρόγραμματος για την περίοδο 7-13. Αυτό θα μας απασχολήσει. Έχουμε δει στην επίσκεψή μας επίσης 7 έργα προτεραιότητας, ε, τα οποία θα συζητήσουμε και θα μιλήσουμε και για τις ε, δυνατότητες για την Ελλάδα. Και θα πρέπει σίγουρα να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση, θα συνεχιστεί και αύριο βέβαια αλλά σε μια άλλη κατεύθυνση. Θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση, θα έχουμε και την Επιτροπή Κρέτσου για την απαλλαγή και βέβαια επ' ευκαιρία της ειδικής έκθεσης ε, του Φεβρουαρίου 2016. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους Θα προσπαθήσουμε και εμείς ε, να ε, βοηθήσουμε όσο μπορούμε και ελπίζουμε και εσείς να βρείτε χρήσιμη τη δική μας δουλειά. Θα τα πούμε αύριο σε 9. Καλό απόγευμα.